Sehr geehrte Damen und äh, Κυρίες και κύριοι, σας ε, καλωσορίζω και πάλι τώρα το απόγευμα στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά και τους προσκεκλημένους μας ε, στο στην ημερίδα ε, για τη διάσταση των φύλων στην εμπορία ανθρώπων. και την Μαρία Σοράγια Ράμο. Ράμος, ε, την εισηγήτριά μα Θα ήθελα να καλέσω πρώτη να πάρει το λόγο. Και σύντομα, δεν βλέπω ακόμα να έχει καταφτάσει, τον ε, κύριο Λόπες Αγγιλάρ. Διότι πρόκειται για κοινή ημερίδα, όπου συμμετέχουν και οι δύο εισηγητές και από τη ΦΑΜ και από τη ΛΥΜΠΕ. Τώρα λοιπόν το απόγευμα έχουμε τρεις προσκεκλημένους. Ε, θα ήθελα να τους ε, χαιρετήσω στη σειρά που θα μας παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους. Ε, καταρχάς την κυρία Σίλβια Γουάλμπιοβέ που είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας και διευθύντρια του σχετικού κέντρου στο Πανεπιστήμιο της πόλης του Λονδίνου, την Σούση Χάχεμαν που είναι ερευνήτρια στο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, ασχολείται και με την ε, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την ε, κυρία Λουκρέσια Ρούμπιο Ρεντέλ που είναι διευθυντήρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου στην ε, Φλωρεντία. Θα ακούσουμε πρώτα τις εισηγήσεις σας και σας παρακαλώ ήδη εκ των προτέρων να μην μιλήσετε υπερβολικά γρήγορα, λέει η Πρόεδρος, για να προλαβαίνουν οι διερμηνείς να κάνουν τη δουλειά τους. Και κατόπιν, ως συνήθως, θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων και με τους εισηγητές και με ε, τους ευρωβουλευτές. Κυρία Βάλμπη, σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω για τη διάσταση των φύλων στην ε, εμπορία ανθρώπων. Μιλώ επειδή είμαι ερευνήτρια στον συγκεκριμένο τομέα και ε, έχω συντάξει διάφορες εκθέσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, το, ε, και τη μονάδα που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων. Και ε, μία από τις εκθέσεις αυτές ασχολείται ακριβώς με τη διάσταση των δύο φύλων και ε, έχουμε εκπονήσει και ε, εκθέσεις για την αναθεώρηση της πολιτικής στις προσπάθειες καταπολέμησης του φαινομένου, καθώς και τη συλλογή δεδομένων για την εμπορία ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, και με βάση ε, αυτών, ε, αυτές τις έρευνες θα σας κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη διάσταση των φύλων ε, στην εμπορία ανθρώπων. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για τη διάσταση των φύλων. Μιλάμε καταρχάς για το γεγονός ότι έχει σημασία το φύλο και μάλιστα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα επικαλείται την ε, ίση μεταχείριση και θα αναφερθώ σε αυτή την αρχή όσον αφορά την ε, ιδιαιτερότητα των ε, δύο φύλων. Αλλά Πάμε και πιο πέρα. Εμπειρογνωσία όσον αφορά τα δύο φύλλα, ισορροπία των δύο φύλων στη λήψη αποφάσεων και προχωρώντας πέρα από το επίπεδο ατόμων, προχωράμε σε θεσμούς δημιουργούμε μια ε, θεωρία πρόληψης ε, και εξετάζουμε και την ε, σχέση ανάμεσα στους διάφορους φορείς, ειδικά όπου μιλάμε για πορνεία, για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών και εξετάζουμε τους διάφορους τρόπους που εξετάζουμε το φύλλο στους τομείς αυτούς. Ο πιο απλός ε, τρόπος ε, έχει να κάνει με τον τρόπο που παρέχεται βοήθεια στα θύματα. Τα θύματα είναι δυσανάλογα, σε δυσανάλογο βαθμό ε, γυναίκες και αυτό φαίνεται πιο αναλυτικά στην έκθεση για την ε, συλλογή δεδομένων αλλά και στις περισσότερες άλλες εκθέσεις. Η πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες και κορίτσια, 75% για την ακρίβεια. Η αναλογία γυναικών ε, ε, κυμαίνεται ανάλογα με το είδος εκμετάλλευσης. Όταν μιλάμε λοιπόν για σεξουαλική εκμετάλλευση, η μεγάλη πλειοψηφία, το 95% ε, των θυμάτων, είναι γυναίκες και κορίτσια. Όταν μιλάμε για εκμετάλλευση άλλων ειδών, η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι μικρότερη. 70% ε, όταν μιλάμε για ε, εκμετάλλευση εργατικού δυναμικού και 50% όταν μιλάμε για άλλες μορφές εκμετάλλευσης. Όταν μιλάμε λοιπόν ε, για, την, για τα δύο φύλλα στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων, σημαντικό είναι να εξετάσουμε το είδος της εκμετάλλευσης. Οι διάφορες μορφές εμπορίας ανθρώπων οδηγούν σε διαφορετικές ομάδες θυμάτων ανάλογα με το είδος ε, εκμετάλλευσης. Άλλα είδη εκμετάλλευσης οδηγούν σε άλλες ανάγκες όσον αφορά τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Στην παροχή υπηρεσιών ε, πρέπει λοιπόν να εξετάζουμε το φύλλο και όχι μόνο να εξετάζουμε εάν πρόκειται για άντρε ή γυναίκε, αλλά να εξετάζουμε και τη συγκεκριμένη μορφή εκμετάλλευση. Σεξουαλική εκμετάλλευση απαιτεί άλλα πράγματα από την εκμετάλλευση εργατικού δυναμικού. Είχαμε διάφορε συστάσει. Δεν ξέρω αν διαβάζετε εδώ τα μικρά γράμματα στη διαφάνεια. Αλλιώ ε, θα βρείτε τι πληροφορίε ε, στην έκθεσή μα. Το πιο απλό λοιπόν θέμα είναι να εξετάσουμε τις ε, ανάγκες των θυμάτων ε, που έχουν να κάνουν με το φίλο τους. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είναι άντρες ή γυναίκες, αλλά έχει να κάνει και με τη μορφή εκμετάλλευσης ε, που υφίστανται. Το φύλλο σχετίζεται και με θέματα επιβολής του νόμου οι φορείς επιβολής του νόμου, οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου έχουν επαρκή κατάρτιση, ε, είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τα θέματα των φύλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 10 όργανα, που, 10 ε, οργανισμούς ε, που συντονίζουν τη σχέση με τις αρχές επιβολής του νόμου σε θέματα εμπορίας ανθρώπων. Και περνάνε αυτή τη στιγμή μια διαδικασία ευαισθητοποίησης, έτσι βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα ω προς το θέμα αυτό. Μπορείτε να δείτε τα εγχειρίδια, θα διαπιστώσετε ότι κάποιοι από τους οργανισμούς έχουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα των δύο φύλων από ό,τι άλλοι. Πρόκειται για συνεχιζόμενες προσπάθειες, ε, κάτι που βλέπουμε και στην βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα επιβολής του νόμου οι συστάσεις μας εδώ δόθηκαν για να ληφθεί η υπόψη η διάσταση των δύο φύλων στις καταρτήσεις που συντονίζουν οι διάφοροι οργανισμοί αυτοί. Υπάρχουν σημάδια προόδου, παρόλα αυτά συνεχίζονται οι προσπάθειες. Πιο πολύπλοκο είναι το ευρύτερο θέμα της πρόληψης. Δηλαδή, όχι την άμεση ε, βοήθεια που παρέχεται στα θύματα ή το πώς θα γίνει η δίωξη των ε, εγκληματιών, των διακινητών, ε, είναι το ευρύτερο θέμα του πώς μπορούμε να αποτρέψουμε, να προλάβουμε την εμπορία. Και αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τους ίδιους οργανισμούς και πώς αντιμετωπίζουν τα δύο φύλλα όταν ε, γίνεται η εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, το θέμα που αφορά κυρίως τις γυναίκες, ε, εξετάζουμε ε, το πώς λαμβάνονται υπόψη τα δύο φύλλα στην νομοθετική ρύθμιση. Μερικές φορές η ανάλυση αυτή περιορίζεται σε θέματα προσφοράς και ζήτησης. Πιστεύουμε όμως με βάση τις έρευνές μας ότι το θέμα είναι πιο πολύπλοκο από αυτό δεν υπάρχουν ε, δύο πλευρές μόνο, αλλά τρεις τομείς ε, που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση. Νομοθέτηση ε, σχετικά με την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών, το δεύτερον το κέρδος που αποκτούν τρίτη και την πτυχή αυτού που αγοράζει τέτοιες υπηρεσίες και είναι τρία διαφορετικά θέματα και πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει πολύ διαφορετική πολιτική ε, στο θέμα αυτό από τι Ηνωμένε Πολιτείε, από όπου προέρχεται όμως ο μεγαλύτερος όγκος ε, της σχετικής φιλολογίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών σε αντίθεση με τις Ηνωμένε Πολιτείε και αυτό οδηγεί σε σημαντικές διαφορές σχετικά με την ποινικοποίηση και αποποινικοποίηση διότι πρέπει να εξετάσουμε τρεις διαφορές πτυχές που νομοθετούνται, που ρυθμίζονται νομοθετικά. Παροχή υπηρεσιών, ε, το κέρδος τρίτων ε, και την ε, αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα προσφοράς και ζήτησης, πρέπει να το εξετάσουμε ως τρίγωνο. Και Το επίκεντρο εδώ είναι στους τρίτους που κερδίζουν, δηλαδή όχι το θύμα της ε, εμπορίας, ούτε ο αγοραστής των υπηρεσιών. Αλλά αυτός που βάζει τα χρήματα στην τσέπη του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ποινικοποιεί αυτήν την πτυχή και στον τομέα αυτών έχουν γίνει τα περισσότερα πειράματα στα κράτη-μέλη. Έχουμε ε, μελέτες από τη Γερμανία, τις κάτω χώρες και την Σουηδία και όπως βλέπετε στην διαφάνεια υπάρχουν διάφορες ε, σχέσεις ε, στις προσπάθειες νομοθετικής ρύθμισης του τομέα αυτού ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε την εμπορία ανθρώπων σε αυτόν τον πολύπλοκο τομέα ανταλλαγών θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην πολυπλοκότητα του θέματος αυτού. Να μην ε, απλουστεύουμε την συζήτηση υπερβολικά στο αν θα ποινικοποιήσουμε ή αποποινικοποιήσουμε συγκεκριμένες πράξεις. Οι καινοτομίες που πραγματοποιούνται στόχο είχαν να μειώσουν την ζήτηση υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας. Η συμβατική προσέγγιση ήταν να επικεντρωνόμαστε πολύ στενά στα θύματα Ε, ή ε, τους εγκληματίες. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη οπτική, να λάβουμε υπόψη μας όλους τους φορείς και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στους τρίτους που κερδίζουν από τις συναλλαγές αυτές. Που αποτελεί ξεχωριστό τομέα νομοθεσίας από αυτόν που αφορά την πώληση και αγορά ε, την παροχή και αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. Οι περιπτώσεις που εξετάσαμε από τις κάτω χώρες και τη Γερμανία έδειξαν πολύπλοκες εξελίξεις. Ε, θεωρούνται εν μέρη τόποι ε, του κέρδους από τρίτους, αλλά η αποποινικοποίηση αυτή και η απελευθέρωση δεν ήταν ε, απλές πράξεις, ενώ είδαμε εν μέρη αποποινικοποίηση της κερδοσκοπίας από τρίτους, ε, είδαμε σημαντική αύξηση προσπαθειών ε, ε, ρύθμισης ε, που προσπαθεί να περιορίσει τα εγκληματικά στοιχεία στην εμπορία ανθρώπων. Με επιτυχία ή όχι, αυτό είναι το ερώτημα. Τα στοιχεία, τα δεδομένα που, στα οποία βασίζεται αυτή η ανάλυση είναι λιγότερο σαφή από ότι οι άλλες πανεπιστημιακές μελέτες. Οι συστάσεις που κάνουμε εδώ πέρα λοιπόν αφορούν τη βελτίωση της συγκέντρωσης δεδομένων, διότι χρειαζόμαστε πιο ε, δυνατή βάση για τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα αυτών. Τα ενδιάμεσά μας συμπεράσματα ήταν καταρχάς ότι πρέπει να ε, επικεντρωθούμε στην πολυπλοκότητα της ε, ρύθμισης που γίνεται, αλλά επίσης στις χώρες αυτές δεν ίσχυε ότι είχε ομαλοποιηθεί η εργασία ε, στον τομέα παροχής σεξουαλικής, σεξουαλικών υπηρεσιών. διότι ε, ακόμα και στις χώρες ε, που είχαν προχωρήσει περισσότερο στην ε, ομαλοποίηση της της, της, στη ρύθμιση του τομέα αυτού διαπιστώσαμε ότι δεν είχε ομαλοποιηθεί τελείως η κατάσταση. Η σουηδική μελέτη έδειξε ότι Ε, είχαμε χαμηλότερα ποσοστά όσον αφορά την ε, εκμετάλλευση ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά ε, αμφισβητούνται τα δεδομένα. Η σουηδική μελέτη έδειξε ότι υπήρχε λιγότερη εμπορία και λιγότερη παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών, αλλά τα δεδομένα δεν ήταν αδιαμφισβήτητα. Έχουμε λοιπόν κάποιες συστάσεις για το πώς θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες και έχουμε και κάποιες προειδοποιήσεις. Πρέπει να βελτιωθούν τα δεδομένα, πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για την τυποποίηση των δεδομένων, ώστε να είναι συγκρίσιμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι τρόποι μέτρησης και εκτίμησης ε, και περνώ στα συμπεράσματά μας. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η πολυπλοκότητα της ε, νομοθετικής ρύθμισης του τομέα παροχής ε, σεξουαλικών υπηρεσιών ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη το πιο προηγμένο σύστημα ρύθμισης στον κόσμο. Είναι πολύ διαφορετικά οργανωμένη η ρύθμιση από τις Ηνωμένε Πολιτείες και έτσι ε, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε εδώ, ε, τα, δεν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ τη συζήτηση περί, απο, που πραγματοποιείται στις ΗΠΑ. Ε, είναι πολύ πιο εκλεπτισμένη η νομοθετική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τέτοιες δραστηριότητες. Θα πρέπει να εξετάσουμε τους διάφορους φορείς ε, και να μην περιοριστούμε στην ε, βοήθεια προς άτομα ή την δίωξη ατόμων. Πρέπει να εξετάσουμε τους φορείς που θα πρέπει να εξετάσουμε στη συνέχεια και επικροτούμε τις προσπάθειες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, προώθηση περαιτέρω μέτρων σε μια ήδη επιτυχή προσέγγιση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτού δώσω το λόγο στην επόμενη προσκεκλημένη μας, ε, θα ήθελα να πω ότι θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε την σειρά, διότι ο συνεισηγητής μας, ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ, ε, δεν θα μπορέσει να παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της ακρόασης. Θα ήθελα λοιπόν να διακόψω, να δώσω το λόγο στον Χουάν Φερνάντο Λόπες και κατόπιν ε, στην συνεισηγήτρια για να μας παρουσιάσουν μια επισκόπηση για να συνεχίσουμε κατόπιν με την ακρόασή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση τη συνεργασία και ευχαριστώ πολύ τη Σωράγια γιατί πραγματικά δυστυχώς έτσι γίνεται στο Κοινοβούλιο. Ε, φοράμε διάφορα καπέλα, έχουμε διάφορες υποχρεώσεις ε, και ε, σε λίγο θα πρέπει να μιλήσω σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά αλλά ταυτόχρονα. Πολύ διεξοδική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όσο και ε, ε, ευαίσθητη αυτή η παρουσίαση, το θέμα της δηλαδή. Εμείς ε, ήδη από το 2016 είχαμε αποφανθεί ότι αυτή, αυτό το εργαλείο για τη βοήθεια των θυμάτων είναι ε, πραγματικά το καλύτερο εργαλείο για την ε, καταπολέμηση του τράφικινγκ και αυτή της διάστασης φύλου. Και βεβαίως ε, καλούμε τα κράτη-μέλη να πάρουν εξειδικευμένα αναφύλο μέτρα και εγώ ίδιος, αλλά φαντάζομαι και η συνεισηγήτρια της ε, ΦΑΜ, ε, θέλουμε implementation report ε, για το θέμα αυτό και εγώ είμαι εισηγητής γι' αυτό και θέλω, έχω σαφώς την πρόθεση να επικεντρωθώ ε, σε προβλήματα ελλείψης, ε, εξέταση όλων των θεμάτων έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η προστασία των θυμάτων που έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, ως θύματα τράφικινγκ, ειδικά για θύματα τα οποία έχουν υποστεί βία. Ε, είναι όντως όπως ακούσαμε και πριν στην προηγούμενη, στην έκθεση που μόλις ακούσαμε ότι πάνω από 60% των γυναικών, των θυμάτων τράφικινγκ είναι ε, γυναίκες και κορίτσια. Αυτό φαίνεται και στην έκθεση του 16. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ε, ε, συγκεκριμένες απαντήσεις. Επίσης ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχυνθεί η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας. Εμείς διαρκώς συζητούμε όχι για τη νέα νομοθεσία αλλά και για την πλήρη εφαρμογή των νομοθεσιών από τις χώρες. Αυτό θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σε αυτήν την ε, οδηγία, λαμβάνοντα υπόψη το ευάλωτο ε, των ε, γυναικών, αλλά και συγκεκριμένων ομάδων, όπως είναι οι ετούντες άσυλο, μετανάστες κλπ. Επομένως, ε, θα πρέπει να έχουμε ένα συντονισμένο και συνεχτικό πλαίσιο ε, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες, τις εξειδικευμένες ανάγκες των ειδικών ομάδων ε, θυμάτων ε, γυναίκες, κορίτσια, τα κορίτσια που είναι πραγματικά ένα, ε, από, ένας από τους πρώτους στόχους ε, της οδηγίας για τα θύματα. Επίσης, να καταπολεμήσουμε τη λαθρεμπορία μεταναστών, γιατί από αυτό τον πληθυσμό των διακινούμενων από διακινητές μετανάστες βρίσκουμε πολλά υποψήφια θύματα τράφικινγκ. Ε, το πρόβλημα, η πρόκληση η μεγάλη του μεταναστευτικού ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Ξέρουμε ότι πάρα πολλά είναι τα κορίτσια, οι νέες γυναίκες που διακινούνται για λόγους παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών και διασχίζουν την Μεσόγειο. Επίσης έχουμε παιδιά τα οποία είναι θύματα τράφικινγκ. to Τέταρτον, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία. Γυναίκες, παιδιά, κορίτσια θα πρέπει να μπουν σε αυτήν την ε, συζήτηση, σε αυτήν την εξίσωση. και να μην λησμονούμε ότι η αυξανόμενη ζήτηση από πλευρά των κρατών ε, είναι ένα κύριο ζήτημα, άρα θα πρέπει να ε, πολεμήσουμε, να χτυπήσουμε την ατιμορρησία. Ναι, βεβαίως, γιατί είναι προφανές ε, ότι Μερικές φορές προστατεύουμε τα θύματα σαν να ήταν ε, θύματα μίας ε, ε, αδύνατον να αποφευχθεί κατάστασης, σαν να ήταν θύματα της μοίρας. Όχι, εδώ έχουμε ποινικέ διαδικασίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταναλώνουν τις ε, σεξουαλικές ε, υπηρεσίες. Μιλάμε για ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιο είναι το δίκτυο εκμετάλλευσης το οποίο κρύβεται πίσω από αυτήν την σεξουαλική υπηρεσία. Επομένως, ναι, το θέμα είναι ευαίσθητο, θα πρέπει οπωσδήποτε όμως να αντιμετωπιστεί. 5. Ε, διασυνοριακή συνεργασία των δυνάμεων καταστολής, εφαρμογής του νόμου, αλλά και δικαστικής συνεργασίας, έτσι ώστε ε, να αποφύγουμε το λεγόμενο forum shopping. Ε, αυτό δηλαδή που προσπαθούν όλοι να βρουν την χώρα με το ευνοϊκότερο καθεστώς. Έκτο, θα πρέπει να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο για, για το trafficking με, με, με ε, σημεία σύγκρισης, benchmarks, καθώς επίσης ε, και σαφή τρόπο αντιμετώπισης της νομοθεσίας ε, και του τρόπου με τον οποίο οδηγούμαστε στην νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στην Μαρία Σοράγια Ροδρίγες Ράμος που είναι η συνεισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τις εμπειρογνώμονες ε, οι οποίες ε, μας συνοδεύουν εδώ. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι θα μας βοηθήσουν και τον Χουάν Φερνάντο και εμένα την ίδια, την, στην Επιτροπή Λίμπε και την Επιτροπή ε, ΦΑΜ έτσι ώστε να μπορέσουμε εν τέλει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εστίαση στην έκθεση που ετοιμάζουμε για την, με την ευκαιρία του νομοθετήματος της οδηγίας για το τράφικινγκ. Όπως είπε και ο Χουάν Φερνάντο προηγουμένως, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε την ε, μεταφορά και την υλοποίηση, ε, την βέλτιστη δυνατή ε, υλοποίηση ε, το, από την πλευρά των κρατών μελών. Μιλάμε για τα εργαλεία τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία μπορεί να έχει η, Επιτροπή ε, στην διάθεσή της, αλλά και τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας εμείς, τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, πολεμήσουμε αυτήν την φοβερή ικτρή κατάσταση του τράφικινγκ. Όπως έλεγε ο Χων Φερνάντο προηγουμένως, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε και πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το φαινόμενο του τράφικινγκ και πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε από τη σκοπιά της έμφυλης διαφοράς, της διάστασης του φύλου. στο τράφικινγκ ε, ανθρωπίνων ε, ειδών, το μεγαλύτερο ανθρώπων, το μεγαλύτερο κομμάτι, 90% αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση και 90% από αυτών των ε, ανθρώπων που είναι θύματα εκμετάλλευσης είναι νέες γυναίκες, γυναίκες και, και κορίτσια. Άρα η διάσταση του φύλου είναι ήδη πολύ σημαντική. Το 1 τέταρτο των, του τράφικινγκ ε, αφορά το, ε, την εργασιακή εκμετάλλευση σε διάφορους τομείς και σε διάφορα ε, πλαίσια σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και από την, το, την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. και 35% ε, είναι ε, αγόρια, άνδρες, ενώ το 75% ακόμα και στην εργασιακή εκμετάλλευση είναι κορίτσια και γυναίκες ε, που τις εκμεταλλεύονται με σαν οικιακές βοηθούς κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε ακριβώς την προσοχή μας σε αυτήν την έκθεση υλοποίηση, οπωσδήποτε από τη σκοπιά της προστασίας των θυμάτων, αλλά οπωσδήποτε ε, και για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας ε, οι εγκληματίες, αυτοί οι οποίοι ε, εμπίπτουν σε αυτό το ποινικό αδίκημα του τράφικινγκ χρησιμοποιούν μηχανισμούς συγκεκριμένους για να διαπράξουν αυτά τα εγκλήματα ε, και οι εγκληματίες ε, ε, τροποποιούν διαρκώς τη μεθοδολογία εργασίας τους χρησιμοποιούν λιγότερο την φυσική βία αλλά χρησιμοποιούν περισσότερο την συναισθηματική βία, την ψυχολογική βία καθώς επίσης και τις νέες μορφές μέσω ίντερνετ, κοινωνικών δικτύων κλπ. Επίσης, ε, συνεργάζονται με διασυνοριακό τρόπο, ε, διαθέτουν μονάδες ε, σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στις χώρες στις οποίες καταφθάνουν εν τέλει τα θύματα του τράφικινγκ, αλλά και στις χώρες προέλευσης των θυμάτων και στις χώρες τράνζιτ, διαμετακόμισης, διέλευσης. Επομένως θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία αν θέλουμε αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε το τράφικινγκ. Ε, επομένως διαστηνοριακή συνεργασία, συνεργασία ε, της σε αστυνομικό επίπεδο, σε ε, επίπεδο δικαστικής συνεργασίας. Ξέρουμε και από την Europol και από την Eurojust ότι τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν υπάρχει εν τέλει καλή συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών υπηρεσιών των μελών. Και επίσης οι κοινέ διερευνήσεις ε, οι οποίες μπορεί να δείξουν καλά αποτελέσματα είναι οι ε, οικονομική φύσεως ε, διερευνήσεις. Όταν μιλάμε για τράφικινγκ, ε, και για σεξουαλικές ε, υπηρεσίες, μη λησμονούμε ότι παράγει, ε, παράγουν οι υπηρεσίες αυτές τεράστιο κέρδος. Επομένως, το, η παρακολούθηση της πορείας του χρήματος και η καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος αποτελεί ένα από τα κεντρικά στοιχεία υλοποίησης αυτής της προσπάθειας και επιτυχίας της προσπάθειας. Θα συνεχίσουμε τώρα βέβαια να ακούμε τις εμπειρογνώμονες και έχω να πω το εξής που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου και στη δουλειά που κάνω για αυτήν την έκθεση. Θα πρέπει να έχουμε στοιχεία και θα πρέπει να δουλέψουμε από κοινού έτσι ώστε ε, να έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη ή να μας δίνουν τα κράτη-μέλη ε, καλύτερα στοιχεία, καλύτερης ποιότητας, ε, συνεκτικά μεταξύ τους. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστούν όλα τα θέματα των μητρών που κρατούνται από τις δικαστικές ή αστυνομικέ αρχές, από την αντιμετώπιση που έχουν ένα καλύτερο αρχείο και αρχιοθέτηση των τρόπων τρόπων αντιμετώπισης ε, του τράφικινγκ από πλευράς ε, των κρατών. Ε, άρα θα πρέπει να βελτιωθεί και πολύ μάλιστα η συλλογή των δεδομένων γιατί τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι πολύ καλά, τα δεδομένα που μας δίνουν τα κράτη-μέλη και από την άλλη πλευρά δεν είναι συνεκτικά μεταξύ τους. Όλοι στα κράτη-μέλη γνωρίζουμε ότι τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μας δείχνουν ότι πάνω από το 60-70% ε, το, του τράφικινγκ γίνεται για λόγους σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ότι 80-90% αφορά γυναίκες και ε, ε, παιδιά. Εδώ όμως δεν έχουμε αναλυτική ε, δυνατότητα να δούμε τα στοιχεία. Δεν βλέπουμε δηλαδή και τις ε, διάφορες μορφές ε, εκμετάλλευσης. Μιλάμε γενικά για εκμετάλλευση ενώ Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες όσον αφορά το τράφικινγκ και όσον αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαι δε απολύτως πεπισμένη ότι πέρα από αυτήν την συνάντηση ε, θα έχουμε την δυνατότητα να συνεργαστούμε μαζί σας και αργότερα, κυρίως ε, σε σχέση με κάποια θέματα τα οποία αναφέρατε και τα οποία μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα και τα οποία θα ήθελα να έχουμε αργότερα την δυνατότητα να τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επισκόπηση αυτή, την εισήγηση που μας κάνατε και δίνω τώρα το λόγο στην ε, δεύτερη προσκεκλημένη μας. Παρακαλώ. Yes. Thank you so much, first of all. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Πολύ ενδιαφέρον και για εμάς να έχουμε αυτόν τον διάλογο και ανταλλαγή στοιχείων. Να σας μιλήσω λίγο για τις κάτω χώρες και ένα χαρτιστικό παράδειγμα που έχουμε στην υπόθεση της εμπορίας ανθρώπων και επίσης όσον αφορά τα στοιχεία μας ε, αυτά που τα ανέφερε και η κυρία Ράμος για το τι πολιτική μπορεί να έχουμε τεκμηριωμένη με στοιχεία και τι άλλο μπορεί να γίνει ε, ονομάζομαι Σουζ Χάχεμαν και ασχολούμαι με αυτή την ε, ε, δουλεμπορία ανθρώπων και είμαι η συγγήτρια πάνω σε αυτό και τη σεξουαλική βία. Ήδη από το 2000 υπήρχε αυτή η θέση, αλλά το 2013 όμως είχαμε την νομοθετική σχετική κάλυψη. Και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από τη θέση μου είναι ότι πρόκειται για ανεξάρτητο φορέα, ανεξάρτητη υπηρεσία και αυτό σημαίνει ότι ενώ μας δίνει κάποιες αρμοδιότητες ο νόμος απει αξιοποίηση αυτών των αρμοδιοτήτων η άσκησή τους ε, κρίνεται το πώς θα γίνει από τον ε, εθνικό εισηγητή. Και οι βασικές αρμοδιότητες μας είναι να μπορούμε για αυτά τα δύο θέματα να κάνουμε έρευνα ε, σεξουαλική βία δηλαδή κατά ανηλίκων και δουλεμπόριο και είπαμε ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαισία του νόμου και συνήθως ε, υποβάλλουμε περιοδικά και κάποιες ε, εκθέσεις και έχουμε και θεματική έρευνα για θέματα που δημιουργούν ανησυχία και προβληματισμό. Τώρα, για να δείτε λίγο τις διαστάσεις του φαινομένου στις κάτω χώρες. Ε, μια εξέλιξη πολύ σημαντική τα τελευταία ένα δύο χρόνια είχαμε και τη σχετική μελέτη αξιολόγησης ότι η τάξη μεγέθους των θυμάτων φέρονται 5 με 7.500 αυτά τα θύματα επειδή το πόσων έχουν καταγραφεί. Αυτό σας δίνει το πλαίσιο της καταστάσεως αλλά δεν έχετε έτσι όλο το τοπίο. Γιατί ξέρουμε, πάντα ξέραμε, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Θα δούμε τώρα σε τι πλαίσιο γίνονται όλα αυτά. Για να δείτε κατά πόσον αυτό είναι απλώς η κορυφή του παγόφωνου. Έχουμε τώρα μια αξιολόγηση πολλαπλών συστημάτων. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες αυτής της μεθόδου, αλλά όποιος θέλει μπορεί να δει αυτή την ε, μελέτη και να έχει όλα τα στοιχεία για το πώς καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Άρα, είπαμε, ετησίως 5 με 7.500 είναι ετησίως τα θύματα ε, αυτού του δουλεμπορίου. Και επίσης, αν με το πόσα θύματα έχουν καταγραφεί, το 2018 ε, έχουμε μόνο 668 καταγεγραμμένα θύματα. Τα βλέπετε αυτά στο δεξί μέρος της οθόνης. Βλέπετε όμως ότι μόνο για την κορυφή του παγόβουνου. Το πόσοι είναι οι καταγεγραμμένοι. Βεβαίως αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εξηγεί το πόσο καλά τα πάμε. Παρ' αυτά όμως παρά είναι μεγάλη αυτή η αριθμή. Και συναντήκαμε με τη Σίλβια, τους συνεισηγητές και συζητήσαμε τι γίνεται. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν η διάκριση του τι είδου ε, ε, παραλλαγές των κλίματος έχουμε. Εδώ μπορείτε να δείτε τους διαφορετικούς τύπους, διαφορετικά είδη δουλεμπορίου και έχουμε το 46% αυτών των θυμάτων που πρόκειται για εκμετάλλευση σεξουαλική στο εσωτερικό της χώρας. Κατόπιν, διασυνοριακά, ε, τα θύματα έρχονται από το εξωτερικό και υφίστανται την εκμετάλλευση στη χώρα μας, 21% και το υπόλοιπο 33% είναι αντικείμενο εκμετάλλευση σε επίπεδο εργασιακό και ποινικό. Αλλά βλέπουμε ότι περισσότεροι είναι ε, προς το θύμα το οφείλονται στη διάπραξη του εγκλήματος στο ιστορικό της χώρας και έτσι αρχίζει κανείς να συνειδητοποιεί το πώς αυτοί οι υπολογισμοί και όσοι προκύπτουν από αυτούς μας οδηγούν στο πού θα δώσουν προτεραιότητα από πλευράς νομοθετικής και πολιτικής γενικότερα επί τη βάση πάντα αυτών των στοιχείων. Άρα μιλούμε για διακίνηση στο ιστορικό, αυτό σημαίνει 3.000 θύματα κάθε χρόνο. Ε, σχεδόν ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι γυναίκες και η, μισή είναι ανήλικοι, ανήλικες. Άρα μιλούμε για Ολλανδέζες. Και αυτοί οι ανήλικοι ε, είναι ακόμα λιγότερο διακριτή. Άρα, πολύ λίγοι δηλαδή από αυτούς τους 1.300 ανήλικους ή ανήλικες έχουν καταγραφεί. Οπότε καλύπτουμε εδώ και ανήλικους και ανηλίκους. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο, γιατί ξέρουμε τώρα πού θα εστιάσουμε την προσοχή μας, σε ποια ομάδα θυμάτων. Για την πρόληψη πρέπει επομένως να κάνουμε δουλειά μέσα από τα σχολεία. Να δούμε πώς θα στοχεύσουμε τις ανήλικες. Είπαμε ότι είναι 1.300 αυτά τα παιδιά ε, φοιτούν σε σχολεία. Αυτό είναι αρκετό κίνητρο επομένως κανείς να ξεκινήσει τη δουλειά με φορείς, με διάφορους εμπλεκόμενους με σκοπό την πρόληψη. Γιατρούς, γονείς, όλοι αυτοί να έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα. Άλλο παραδείγμα τώρα έχουμε το λεμπόριο σε σχέση με το φύλλο των θυμάτων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας για την εκμετάλλευση στο εσωτερικό ε, βλέπετε εδώ το πράσινο χρώμα σχεδόν 100% γυναίκες για αυτή τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Μετά πάμε στο διασωριακό έγκλημα, έχουμε λίγο περισσότερους ε, άνδρες, γύρω στο 18%. Μετά εργασιακή εκμετάλλευση και γενικά ποινικού, ποινικά κολάσιμη εκμετάλλευση. Εδώ έχουμε τους μισούς και πάνω. Άνδρες. Τώρα, όσον αφορά το πόσα θύματα έχουν καταγραφεί, αλλάζουν κάπως τα πράγματα. Ανεβαίνουν τα ποσοστά των γυναικών σε κάθε κατηγορία. Αυτό μας λέει ότι τα θύματα εκμετάλλευσης εργασιακής και διασυνοριακής δεν έχουν καταγραφεί. Σε σχέση τώρα με το σύνολο, κανείς βλέπει τις διαστάσεις του θέματος. Δεν αναφέρονται όλα τα Άρα ένα θύμα το για την σεξουαλική εκμετάλλευση αλλά και όσον αφορά τα εργασιακά ίσως θα πρέπει να εξετάσουν περισσότερους ε, κλάδους, τομείς της οικονομίας. Που σε ποιες δουλειές, που έχουν περισσότερες γυναίκες και έτσι καταλαβαίνετε το πλαίσιο. και επίσης αυτά είναι στοιχεία που τροφοδοτούν την Eurostat. Είναι χρήσιμα αυτά τα στοιχεία και έτσι διαμορφώνονται το ποιες προτεραιότητες τάσουμε. Άρα, τώρα ποια είναι τα προβλήματα, οι προκλήσεις όσον αφορά την αξιοποίηση των γεγονότων, των στοιχείων τέλο πάντων, για την πολιτική, το πρώτο θέμα βέβαια είναι η αξιοπιστία των στατιστικών, δεν τα πάμε άσχημα στην Ευρώπη όσον αφορά την συλλογή των στοιχείων. Πρώτα-πρώτα το θέμα είναι η νομοθεσία για προστασία ιδιωτικού βίου για την καταγραφή των θυμάτων, πληροφορίες, προσωπικών στοιχείων Άρα, συλλογή στοιχείων και ταυτόχρονα προστασία του ειδικού βίου των θυμάτων. Σε αυτό είναι πιο εύκολη δουλειά της αστυνομίας. Μπορούν να μας αναφέρουν πιο ελεύθερα το τι γίνεται. Όμως ε, για τα πιο νέα θύματα του δουλεμπορίου δεν εμποδίζει την καταγραφή η νομοθεσία για προστασία ιδιωτικού βίου. Οπότε έχει πρόβλημα και η αστυνομία σε αυτό. Ε, πολλές φορές ε, έχουμε και θέματα σχετικά με το μεταναστευτικό. Το ίδιο το μεθοδευτικό είναι πρόβλημα και άρα το ζήτημα το τι προτεραιότητα έχει η αστυνομία. Ίσως δεν ασχολούνται αρκετοί και να υπάρχει μια σφαιρική άποψη του τι γίνεται σε σχολεία, ε, οι γιατροί πολλές φορές πιο κοντά στα θύματα είναι οι δημοτικές, κοινοτικές αρχές άλλο πρόβλημα ότι αυτά τα δεδομένα δεν μας δίνουν το σύνολο του τοπίου. Γιατί όσον αφορά τους υπολογισμούς βασιζόμαστε στη διαχρονική καταγραφή. Σύμφωνοι, καλό αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποια νέα φαινόμενα που δεν τα γνώριζαν προηγουμένως και ε, θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα νέα φαινόμενα να μην πέσουμε στον φαύλο κύκλο του να εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στο τι βρίσκουμε την έρευνά μας. Οπότε το ζήτημα είναι εδώ τώρα για τους ανήλικους που υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση. Ε, εδώ έχουμε και θέματα ναρκωτικών. Κάποιοι από αυτούς είναι λοάδικοι, δεν μπορούν πια να μείνουν στην οικογένειά τους. Έχουμε, είχαμε και μια οργάνωση που εκμεταλλευόταν εκατοντάδες τέτοιους ανηλίκους, ε, δύο ήταν οι εν προκειμένου, και να δούμε πόσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και αυτό εξηγεί γιατί δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ε, στη μελέτη μας γιατί κανείς δεν τα καταγγέλει, δεν τα αναφέρει. Τώρα, εκμετάλλευση εγκληματικού χαρακτήρα, πολλές φορές αυτή είναι Ρώμα, Βιετναμέζοι κυκλώματα ναρκωτικών. Αλλά δεν αναφέρονται καθόλου Ολλανδία. Αλλά γνωρίζουμε όμως από γειτονικέ χώρες ότι έχουμε εδώ πάρα πολύ σοβαρά εγκλήματα νέοι άνθρωποι τα κάνουν και επιστρατεύονται πολλές φορές εξαναγκάζονται τα θύματα να προβούν σε εγκληματικές ενέργειες. Αλλά θα πρέπει να τα βλέπουμε από τη σωστή οπτική γωνία. Όπως είπαν οι συνειζηγήτριες, έχουμε το ζήτημα της ε, μετανάστευσης μεγάλης κλίμακας. Προβληματικό αυτό, γιατί αν βλέπουμε τα στοιχεία και τα συγκρίνουμε για όλη την Ευρώπη, ε, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε το φαινόμενο και για κάθε έγκλημα που θα καταγραφεί ε, το θύμα. Αν κάτι γίνει, ε, αν το έγκλημα γίνει καθοδόν προς την Ολλανδία θα το καταγράψουν οι Ολλανδοί. Αλλά μπορεί να έχει περάσει πριν το θύμα από την Ιταλία. Πού θα καταγραφεί, πού θεωρείτε ότι έγινε η εκμετάλλευση. Φυσικά και πρόκειται περί ευάλωτων προσώπων, Οπότε αυτό εκμεταλλεύονται εις βάρος του θύματος και αυτό για την προλήψη πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και αυτό θα πρέπει να είναι και το κλειδί για το ζήτημα αυτό. σημαντικό πρόβλημα εδώ είναι για τιμωρησία που γίνεται. Πολλές φορές κάποιος με τιμωρητός και αυτό αφορά πολλά θύματα, άρα θα πρέπει να εξετάσουμε για την πρόληψη και το τι θα γίνεται με τους παραβάτες, με τους εγκληματίες. Δεν έχει γίνει αρκετή έρευνα επίσης σε σχέση με το ποιο και πώς θα πάει να γίνει διακινητής, λαθροδιακινητής μάλλον. Και αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος. Είμαι κάπως πιο ευέλικτη σήμερα, διότι ξέρω ότι κάποιοι πρέπει να φύγουν, άλλοι προσέρχονται. Ε, ζητώ την κατανόησή σας. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην Francis Fitzgerald. Πρωτού προχωρήσουμε στην ε, επόμενη παρουσίαση, διότι ε, πρέπει να αποχωρήσει. Και κατόπιν θα φτάσουμε στην τρίτη παρουσίαση και θα συγκεντρώσουμε όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, το εκτιμώ αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο μιλήτριες για ε, τις μελέτες τους ε, που νομίζω ότι θα είναι πολύ ε, χρήσιμες για την, για εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Απομένουν πολλά να γίνουν στο θέμα αυτό. Τώρα ανοίγει η αυλαία. Η σχετική νομοθεσία αναθεωρείται αυτή τη στιγμή και συχνά γίνεται προσπάθεια υπονόμευσης της νομοθεσίας. Θα... Ήθελα να πω ότι εμένα με παρεξενεύει ότι δεν υπάρχει ακόμη περισσότερη οργή για το θέμα αυτό στα κράτη-μέλη από ό,τι βλέπουμε, διότι είναι κάτι το οποίο ε, πληγώνει πάρα πολύ τις ε, γυναίκες ε, που πέφτουν θύμα της εμπορίας ανθρώπων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουμε εδώ. Κάτι θα ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά τη διάσταση των δύο φίλων σε σχέση με τους ε, φορείς της δικαιοσύνης. Ε, συνήθως αυτοί δεσπόζονται κυρίως από άντρες ε, και είτε μιλάμε για τον Frontex, τον Europol ή άλλους οργανισμούς, απομένει πολλή δουλειά να γίνει στον τομέα της δικαιοσύνης όσον αφορά την κατάρτιση σε θέματα ε, διάστασης των ε, δύο φύλων. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό, διότι είναι κάτι απολύτως απαραίτητο. Όσον αφορά τη δεύτερη μελέτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την έρευνα αυτή. Ε, τίθεται το όλο θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών και το τι γίνεται με ε, τα ανήλικα που περιγράφεται στη μελέτη σας. Το 50% των θυμάτων λέτε ότι είναι κάτω των 18 ετών. Ε, είναι πράγματι συνταρατικά αυτά τα στοιχεία. Χρειάζεται πολύ πιο εντατική αστυνομική δουλειά πάνω στα θέματα αυτά. Είμαι βέβαιη ότι έχετε δίκιο όσον αφορά και τους άντρες και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, και πολλά νέα αγόρια υφίστανται κακοποίηση. Σας ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, πράγματι η κατάρτιση συμβάλλει σημαντικά ε, στην βελτίωση των ε, αρχών επιβολής του νόμου για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Και όχι μόνο κατάρτιση. Άλλη σημαντική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ισορροπία των δύο φύλων ε, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και αναφέρατε πόσοι από τους φορείς αυτοί δεσπόζονται από άντρες. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε περαιτέρω μήπως η ισορροπία των δύο φύλων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που τώρα επεκτείνεται και σε διάφορους άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βλέπουμε για παράδειγμα τη συζήτηση για τα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Μήπως η αρχή αυτή λοιπόν ε, μπορεί να διευρυνθεί και να καλύψει και τους ε, οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη. Θα ήθελα λοιπόν να το προσθέσω και αυτό στον κατάλογό σας. Και τέλος, σε ένα τελευταίο θέμα όσον αφορά την ποινικοποίηση. Η ποινικοποίηση, σύμφωνα με την οδηγία, είναι άνηση και μπορεί να αξίζει το κόπο να το εξερευνήσουμε αυτό περαιτέρω. Δεν έχουμε ποινικοποιήσει αποτελεσματικά όλα τα κράτη-μέλη της πράξης που ε, ε, προτείνει η οδηγία ότι θα μπορούσαν να ποινικοποιηθούν. Και αυτό αποτελεί ίσως ένα στοιχείο που μπορούμε να προσθέσουμε στο πλαίσιο της ε, ισχύουσας οδηγίας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ για την ε, παρατήρησή σας. Ναι, συμφωνώ απολύτως όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών ε, και τα ανήλικα. Ήταν πολύ ανησυχητικό αυτό το στοιχείο που προέκυψε από τη μελέτη. Και ε, οι ερευνητικοί φορείς θα πρέπει όχι μόνο να εξετάσουν το θέμα της κατάρτισης και κάποια από τα άλλα θέματα που αναφέρατε, διότι βλέπουμε ε, τον δισταγμό νέων κοριτσιών να καταγγείλουν ε, ε, τις πράξεις αυτές στην αστυνομία, διότι ταπεινώνονται, βλέπουμε πώς η αστυνομία χειρίζεται τέτοιες αναφορές. Ακούμε, για, ακούμε περιπτώσεις όπου η αστυνομία δεν έχει χειριστεί σωστά το θέμα. ακούμε περιπτώσεις όπου οι γυναίκες έχουν κάνει μήνυση για εμπορία ανθρώπων ή σεξουαλική ε, επίθεση, αλλά είναι ένα θέμα που συνδέεται ήδη με την ε, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Από πολύ μικρά θα πρέπει τα αγόρια και τα κορίτσια να μαθαίνουν ε, πώς να συναναστρέφονται μεταξύ τους διότι ε, τα θύματα θα πρέπει να καταλαβαίνουν ότι αυτό που τους συμβαίνει είναι λάθος, είναι κακό και τους δίνει έτσι περισσότερο θάρρος ώστε να πάνε να καταγγείλουν τις περιπτώσεις αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στην επόμενη ομιλήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να παρουσιάσω την έρευνά μου εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία αφορά ε, το θέμα μας. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα ξεκινήσω αμέσως με την παρουσίασή μου θα είμαι σύντομη, δεν ξέρω αν είναι έτοιμο και το powerpoint που πρέπει να δείξω, έτσι ώστε μετά λέω θα είμαι σύντομη για να μπορέσουμε να κάνουμε μετά ε, την, ε, να έχουμε τη δυνατότητα για συζήτηση. Ε, εγώ θα συζητήσω για το θέμα της διάστασης φύλου στις πολιτικές κατά του τράφικινγκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι η εστίαση στο στα θύματα και η ε, διάσταση φύλου. Αυτά είναι δύο θέματα τα οποία σχετίζονται, είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, γιατί αυτοί που θέλουν να πιέσουν ε, να υπάρξει διάσταση φύλου στη, στα μέτρα anti-trafficking ε, είχαν τον στόχο να ξεφύγει από τα όρια το τράφικι, να ξεφύγει από τα όρια της μεταναστευτικής πολιτικής και της, ε, ε, των θυμάτων. Επομένως, στην αρχή της δεκαετίας του 90 ε, και κυρίως μετά από ε, όθηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως της Επιτροπής ε, Γενεκών σε συνεργασία με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών όθησαν έτσι ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές κυρίως αυτές οι οποίες ήθελαν να αντιμετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών. Ε, και ε, για πρώτη φορά δόθηκε διάσταση φύλου ε, σε, αυτές τις, σε αυτά τα αδικήματα γιατί όντως κυρίως αφορούσαν γυναίκες και κυρίως με στόχο την, σεξουαλική, την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών, σεξουαλική εκμετάλλευση. Εδώ είχαμε λοιπόν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών ε, που απέρε από την ε, διάσταση φύλου όσον αφορά αυτές, ε, αυτά τα αδικήματα. Το 2011 είχαμε το επιστέγασμα των προσπαθειών με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βία κατά των γυναικών και τα σχετικά μέτρα και πολιτικές και ξεκίνησε λοιπόν ε, η διάσταση φίλου να ελέγχεται όχι μόνο και να αναφέρεται όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις ε, πράξεις. Οι πολιτικές αντιτράφικινγκ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν το φαινόμενο αυτό το που θίγει ιδιαίτερα τις γυναίκες και επίσης ε, υπήρξαν πολλά μέτρα τα οποία εξέφευγαν ε, τις, ε, των στενών μέτρων ελέγχου των συνόρων κλπ. και οδήγησε σε στενή συνεργασία πολλών υπηρεσιών. Βεβαίως η προστασία ακόμα ελέγχεται από τις γενικότερες πολιτικές μετανάστευσης και καταπολέμησης του τράφικινγκ ε, ωστόσο υπάρχει αυτή η διάσταση ε, των, ε, της διάστασης του φίλου. Βέβαια η μεγάλη επιτυχία ήταν περισσότερο στα λόγια παρά στα έργα. Η απάντηση που βρίσκω για το φαινόμενο αυτό είναι η εξή. Η προσέγγιση της βάση διάστασης φίλου σε σχέση με το τράφικινγκ δεν κατάφεραν να πάρουν τον, δεν κατάφεραν να πάρουν το θέμα αυτό από, την, ε, από το θεματολόγιο της ε, εσωτερικής ε, ασφάλειας και Επομένως, τα μέτρα τα οποία προτείνονται από άποψη διάστασης φύλου δι, ε, ε, συνυπάρχουν και μάλιστα τέμνονται ε, με όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια. Και επομένως έτσι ενισχύεται και διαστέλλεται και η προβληματική αντιμετώπιση, άρα και οι ελλειπείς λύσεις που προτείνονται, γιατί προτείνονται πάντα από την πλευρά της ασφάλειας και όχι από την πλευρά της ε, διάστασης φύλου. Uh, Εάν ε, συγκρίνουμε ε, τα μέτρα για την βία κατά των γυναικών γενικά και τα μέτρα που προτείνονται για την καταπολέμηση του τράφικινγκ προκύπτουν αρκετές διαφορές. Ε, ακριβώς λόγω του ότι τέμνονται ε, τα μέτρα ε, αντιμετώπισης βίας κατά των γυναικών με τα μέτρα για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα το trafficking, βλέπουμε ότι έχουμε περισσότερο μέτρα τα οποία αφορούν την εξωτερική διάσταση, ε, αφορούν δηλαδή ε, ε, και επικεντρώνονται κυρίως στις γυναίκες που είναι θύματα του τράφικινγκ, οι οποίες στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι ξένες γυναίκες. Δεν εστιάζουν τόσο πολύ στο τους, ε, στις προϋποθέσεις ε, που επιτρέπουν ε, την θυματοποίηση και το τράφικινγκ στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν γίνεται μεγάλη εστίαση από την πλευρά της ζήτησης. Ακόμα και όταν όμως αντιμετωπίζεται και το θέμα της ζήτησης, αυτό γίνεται ε, και με αποσυγκεκριμένη οπτική γωνία. Δεν βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει μια στρατηγική επιτυχής. Η δεύτερη διαφορά ανάμεσα στους μηχανισμούς προστασίας ε, που αφορούν ε, γενικά την βία κατά των γυναικών και ε, ειδικά το τράφικινγκ των γυναικών είναι ότι η παρέμβαση περιορίζεται στις πιο ακραίες περιπτώσεις, extreme cases, δηλαδή οπουδήποτε, οποτεδήποτε απειλείται η ζωή του θύματος ή όταν έχουμε ιδιαίτερα υψηλή βία και μεγάλη εν τέλει βλάβη ή όταν μιλάμε για οργανωμένο ε, έγκλημα, δηλαδή όταν ε, αναμειγνύονται οι ε, οργανώσεις του εγκλήματος. Και ίσως η τελευταία αλλά πιο σημαντική διαφορά είναι ότι τα μέτρα τα οποία προστατεύουν τα θύματα του τράφικινγκ βασίζονται στη συνεργασία ε, με τα θύματα και την απόδειξη ότι πραγματικά ε, δεν ε, αποτελούν κίνδυνο ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνεται, προστασία δηλαδή στα θύματα τράφικινγκ αλλά με πολλές προϋποθέσεις συνεργασία, συμμετοχή σε προγράμματα That Προγράμματα επανένταξης ε, κλπ. Ε, δηλαδή τα αφηγήματα των, θυμάτων ε, από την ε, σκοπιά της διάστασης φύλου δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα, την γενικότερη αντιμετώπιση του θέματος της βίας των γυναικών πάντα από την πλευρά της μετανάστευσης, της ε, βίας, του οργανωμένου εγκλήματος, εν τέλει της ασφάλειας. Και επίσης ε, πολλές ε, διεκδικήσεις ε, είναι ας πούμε φεμινιστικού υποβάθρου και χρησιμοποιούνται ε, ευρύτερα νομίζω εγώ ότι θα πρέπει να δούμε την ίδια τη διάσταση του φύλου, να δούμε δηλαδή εάν και κατά πόσον θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν σε αυτήν την συνάντηση με τα μέτρα που αφορούν τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια. Κατά την έννοια αυτή πιστεύω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερη σκέψη, προβληματισμό και ενδεχομένως περαιτέρω βελτίωση. Είναι να καταλάβουμε τη διάσταση φύλου ε, του τράφικινγκ έτσι όπως έχει αντιμετωπιστεί από την αρχή γιατί ε, ε, πραγματικά η διάσταση του φίλου ειδώθηκε πάντα από την σκοπιά της, ε, ε, του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας και προστασίας. Επομένως, ε, βασίζεται πάντα στην, στη, στη βία και την φυσική συναισθηματική βία την οποία έχουν υποστεί, κυρίως σε σχέση με τη μετανάστευση και ε, την ατιμορρησία ε, λόγω οργανωμένου εγκλήματος. In this regard, the possible contradictions that can emerge from the objectives of crime and migration control on the one hand and prevent... Νομίζω ότι εάν δούμε την προστασία των συνόρων και την ασφάλεια από τη μία και την προστασία ε, των θυμάτων από την άλλη, τότε ε, ε, ε, κατανοούμε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί το αδίκημα ή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ο βαθμός της απειλής όταν δεν μιλάμε για νόμιμους μετανάστες. Επίσης ε, υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός μέσω του οποίου ε, η διάστηση του φύλου προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει τις, ε, τα θύματα του τράφικινγκ βάσει του επίπεδου κινδύνου και όχι βάσει της παρανομίας την οποία έχουν ε, υποστεί. Και επομένως εάν υπάρχει ε, κατάχρηση ε, μέσω της τροτότητας ε, ή ακόμα και της σκλαβιάς, της δουλείας. Η έννοια της τροτότητας, vulnerability και της δουλείας slavery λαμβάνονται υπόψη, αλλά όχι όταν μιλάμε για παιδιά. Ε, ελέγχεται δηλαδή ο βαθμός θυματοποίησης αλλά ε, μπορεί να έχει και ε, αντίθετα αποτελέσματα ε, γιατί σε αυτές τις ε, περιπτώσεις ε, η διατομή ανάμεσα στα στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως οδηγούν σε μια αποκλειστική αντιμετώπιση της σκληρότητας ή ενός εξιστασιαλισμού που αφορά μονάχα την αντιμετώπιση της διάστασης του φύλου και επομένως στην ουσία έχουμε δεύτερη θυματοποίηση με τον τρόπο αυτό. Οι έννοιες αυτές έχουν και κάποια ε, δεύτερα, ε, κάποιες δεύτερες επιπτώσεις, γιατί οδηγούν σε μέτρα προστασίας, τα οποία εστιάζουν κυρίως ε, στο ίδιο το τράφικινγκ, συμβάλλουν στον περιορισμό της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πιο ακραίες περιπτώσεις, μέσω της οικοδόμησης ενός αφηγήματος το οποίο περιθεριοποιεί την ε, θυματοποίηση και στην ουσία εν τέλει ε, σχηματοποιεί τα θύματα του τράφικινγκ ως απειλές ε, στην ασφάλεια και την ελευθερία χωρίς να νοιάζονται στην ουσία για την ίδια την ταυτότητα των ε, θυμάτων και σε πολλές περιπτώσεις ε, οδηγούν και τις ίδιες τις γυναίκες να συμμετέχουν σε επικίνδυνες ε, συμπεριφορές. Και επειδή ακριβώς ε, η έλλειψη ελεύθερης βούλησης επιβαρύνεται από την φυσική και ψυχολογική βία, οδηγούμαστε στην διόγκωση του φαινομένου, ενός φαινομένου που όπως είπα και προηγουμένως προκύπτει κυρίως από την διατομή της προστασίας των γυναικών και της ε, ε, βίας κατά των γυναικών, στη διατομή τους λέω, με τον χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Um, in order to correct uh, αυτή η διατομή λοιπόν που είναι εσφαλμένη αντιμετώπιση ε, και που μπορεί να οδηγήσει ε, στο, human, στο, στο trafficking ε, ανθρώπων μας οδηγεί στον συσχετισμό ανάμεσα στην υπετιότητα, την βλάβη, το φύλλο, το τράφικινγκ και την διάσταση φύλου σε σχέση με τη θυματοποίηση και μόνο. Αυτά ήθελα να σας πω. Θα, θα σταματήσω εδώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, λέει η Πρόεδρος. Τώρα δώσουμε τον λόγο στους συναδέλφους. Πρώτη η κυρία Άντερσον. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πολύ πλήρεις παρουσιάσεις, πολλές διάφορες πτυχές ακούσαμε, τις οποίες βρήκα ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρουσες. Αναφέρθηκαν διάφοροι παράγοντες, ε, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφέρω μια άλλη πτυχή. Και εμείς, ως δυτικές κοινωνίες, να το πω έτσι, παρέχουμε ευνοϊκούς παράγονται σε ευνοϊκές συνθήκες για την εμπορία ανθρώπων. Αν μου επιτρέπει η Προεδρία, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Πιστεύω ότι έχουμε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά ε, τις τον τρόπο συζήτησης, την οτροπία στις κοινωνίες μας αναφέρεται η πολιτική ορθότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2002 υποβλήθηκε νέα θομοθεσία στην Γερμανία που στόχο είχε την αποποινικοποίηση της πορνείας. Ε, το επιχείρημα ήταν ότι στιγματίζονται οι γυναίκες και έτσι ε, δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στην αγορά εργασίας. Ε, Οποιοςδήποτε μίλησε κατά της πρότασης αυτής θεωρήθηκε μισογίνης. Ε, αποκλείστηκε ουσιαστικά από τη συζήτηση και ε, η προσέγγιση αυτή ε, υπονοούσε ότι οι γυναίκες από μόνες τους εθελοντικά προχωράνε στην πορνεία. Παραβλέφθηκε τελείως και θυμάμαι πολύ καθαρά τη συζήτηση ήταν αυτό. Αλλά οι γυναίκε δεν το κάνουν αυτό επειδή το θέλουν. Ε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αναγκάζονται ή καταναγκάζονται να το κάνουν αυτό. Είναι λοιπόν θύματα και αποτελούν θύματα εκμετάλλευση Στην Σουηδία είναι τελείω διαφορετική η προσέγγιση. Έχει ποινικοποιηθεί ε, η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. Όποιος ήταν τότε κατά του νέου νομοσχεδίου, ε, αποκλείστηκε από τη δημόσια συζήτηση. Θεωρήθηκε μισογίνης, ε, ε, αντιδραστικός κλπ. Τούτων λεχθέντων, σήμερα όταν συζητάμε το θέμα της εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε όλους τους διαφορετικούς παράγοντες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η πολιτική των ανοιχτών σύνορων σε μεγάλο βαθμό συμβάλλει στο να πέφτουν όλο και περισσότερες γυναίκες θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε σε τι βαθμό βλέπετε εσείς να υπάρχει αυτός παράγοντας και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μην είναι πια τόσο απλό να ε, περνούν ε, ε, διάφοροι άνθρωποι από την Ευρώπη και να καταλήγουν σκλάβοι. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει το λόγο? τότε να ρωτήσω εγώ κάτι. Την καθηγήτρια Βόλμπη. Σε με αυτά που είπατε, τα στοιχεία σας σε σχέση με την Σουηδία. Θα με ενδιέφερε αν μπορείτε να επεκταθείτε για τους Σουηδούς που πάνε στην Γερμανία. Ότι η εθνική νομοθεσία προκαλεί τέτοια αντίδραση. Τι στοιχεία έχετε. Επίσης, Όσον αφορά τους ε, υγειονομικούς ελέγχους, έχετε στοιχεία. Κατόπιν, για την κυρία Χάχημαν. Όσον αφορά την έλλειψη στοιχείων σε σχέση με τις ε, εκθέσεις, τις αναφορές. Αυτό μήπως σχετίζεται με έλλειψη αστυνόμευσης, ε, προβλήματα προσωπικού. Υπάρχει τέτοια σχέση. Έχουν άλλα θέματα προτεραιότητα. Τι γίνεται. Και η Ευχένια έχει όμως ε, κάποια ερώτηση. Η κυρία Παλόπ. Ω, πότε να δώσω το λόγο στην συνεισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τερία θέματα προς τις προσκεκλισμένες μας για να μου πούν αν συμφωνούν με αυτό που με προβληματίζει. Πρώτα-πρώτα, σε αυτές τις περιπτώσεις ε, επικεντρώμαστε στην πλευρά την ποινική αστυνομική. Στην πράξη συχνά τα θύματα δεν έχουν προστασία γιατί δεν δείχνουν οι διοικητικές αρχές ε, την επιμέλεια που χρειάζεται ή δεν θέλουν να συνεργαστούν. Και καταλήγουμε επομένω στο να εξετάσουμε το τι γίνεται όσον αφορά τα σύνορα, τη δημοσία τάξη και τα ποινικά ζητήματα. Οπότε βλέπουμε ότι συνήθως, θυμίζουμε το θέμα του δουλεμπορίου, σε σχέση με την λαθρομετανάστευση. Επίσης, τι γίνεται από πλευράς δικαστικής νομικής. Συνήθως έχουμε αποζημίωση χρηματική, έχουμε ποινική κύρωση και πολλές φορές όμως τα θύματα δεν εισπράττουν την αποζημίωση. επομένω. τι γίνεται σε σχέση με την νομική προστασία και την υποχρέωση του κράτους για προστασία για Επίσης, Είπαμε για εκμετάλλευση εργασιακή σε σχέση με το δουλεμπόριο, ότι όταν αυτά γίνονται εντό συνόρων και την εκμετάλλευση σεξουαλική. Έχουμε εδώ έναν τομέα που είναι από δύο πλευρές Δεν υπάρχει κάλυψη για τα εργασιακά και πολλές φορές κάποιοι προσφέρουν υπηρεσίε κατοίκων, δεν καλύπτονται όπως αλλού, δεν μπορεί να υπάρχει επίσης επιθεώρηση εργασιακή. Για πέστε μου, πώς το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Και τώρα... Μαρία Σοράγια, η συγκεντριά μας. Ευχαριστώ. Για την κυρία Βόλβη. Μα είπες στην εισήγηση για αυτό το τρίγωνο της εκμετάλλευσης όσον αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση και το λεμπόριο. Το τρίγωνο μεταξύ θύματος. Εκμεταλλευτή και του ωφελουμένου, του χρήστη. Ελήφθη υπόψη κατά τη γνώμη σου μία έκθεση της Europol για την δουλεμπορία αυτήν. Λέει εκεί η έκθεση ότι τα κράτη-μέλη που έχουν νόμιμη πορνεία εκεί τι γίνεται με τους ε, ε δουλεμπόρους εκεί διευκολύνεται το έργο τους δυσκολεύεται τα, τα, τα θύματα είναι πιο εύκολο το να απασχολούν τους ε, ανηλίκους και τελικά να καταλήγουν αυτοί σε εκμετάλλευση σεξουαλική. Επίσης έχουμε την οδηγία στο άρθρο 18 και εκεί που έχει την ε, κατάταξη των διαφορετικών υπηρεσιών και μιλάει για αυτούς που ξέρουν ότι έχουν υπηρεσίες ε, από κάποιον που είναι θύμα του δουλεμπορίου. Οπότε εκμεταλλεύονται σεξουαλικά έναν ανήλικο και αυτό γίνεται δολείο, εν γνώση τους. Και βέβαια είναι πολύ πιο αποδοτικό οικονομικά. Για πέστε μας τώρα, τι γίνεται με την εκμετάλλευση στο ιστορικό της χώρας. Το είπε κάποια από εσά. Αυτά λέει και η Κομισιόν στην τελευταία της έκθεση που αφορά το δουλεμπόριο ότι έχει αυξηθεί το δουλεμπόριο εντό των συνόρων τα τελευταία χρόνια και σεξουαλική εκμετάλλευση και εκμετάλλευση για διάφορους σκοπούς ε, εκμετάλλευση εργασιακή, λαθρεμπόριο οργάνων. Για πέστε μου τη γνώμη σα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο για τις ερωτήσεις και τώρα να σας δώσουμε το λόγο για ένα τελευταίο γύρο απαντήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις. Καταρχάς, ε, το μισό της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, έχει να κάνει με τα σύνορα. Μερικοί ε, μιλάνε για εγχώρια εμπορία ανθρώπων. Μόνο το μισό δηλαδή έχει να κάνει με κάποιο σύνορο, τη διέλευση κάποιου σύνορου. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά υπάρχουν κάποια ε, εν μέρη σύνορα και κατόπιν έχουμε τα σύνορα ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τρίτων χωρών. Αλλά επειδή το μισό της εμπορίας δεν έχει να κάνει με διέλευση σύνορων, αυτό αλλάζει την ιδέα των ανθρώπων σχετικά με το τι είναι η εμπορία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περάσει κανείς κάποιο σύνορο. Η εμπορία είναι εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης κάποιου άλλου. Και ενώ τα σύνορα μπορεί να έχουν να κάνουν με την ε, ευάλωτη αυτή θέση, δεν αποτελούν ε, την μόνη αιτία για την ευάλωτη θέση που ε, οδηγεί σε εκμετάλλευση. Είναι απλά ένα παράδειγμα, αλλά δεν είναι η αποκλειστική αιτία για την ευάλωτη θέση. Η δουλειά που κάναμε στη Γερμανία έδειξε ότι κάποιες ε, γερμανικές πόλεις και κομοπόλεις ε, είχαν εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές για να ρυθμίσουν την εμπορία ανθρώπων και την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών. Υπήρχε λοιπόν ε, καινοτόμος τρόπος συνεργασίας ανάμεσα στις κοινωνικές και τις αστυνομικές υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προστάτευσε τους ανθρώπους σε αυτές τις πόλεις, αλλά δεν εμπόδισε την μεταφορά των δραστηριοτήτων αυτών σε άλλες πόλεις σε λιγότερο καλά ρυθμισμένες. Ε, είδαμε λοιπόν τα, στοιχεία αυτά όχι μόνο σε σύγκριση ανάμεσα στη Σουηδία και τη Γερμανία, αλλά είδαμε και εντό τη Γερμανία ε, διαφορά ανάμεσα στις περιοχέ όπου υπήρχε καλή ρύθμιση και στι χώρε όπου δεν υπήρχε. Δύο απαντήσεις δίνονται σε αυτό. Μερικοί λένε αφήστε την ε, νομοθετική ρύθμιση, ενώ άλλοι λένε να είναι πιο συνεπής η νομοθεσία και να μην επιτρέπουμε στην νομοθετική ρύθμιση να αφορά αποκλειστικά μία πόλη εντός μιας χώρας ή μόνο εντός μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες απαντήσεις που δίνονται όσον αφορά τον εκτοπισμό των ε, ανθρώπων, τη, μεταφορά των, ε, τη μετακίνηση των ανθρώπων, ε, αλλά δεν είναι μόνο σημαντική απάντηση. Όσον αφορά το ποινικό δίκαιο, έχουν γίνει διάφορε συζητήσει σχετικά με την νομοθεσία. Εντός της Ευρώπης υπάρχουν διάφορε μορφές νομοθεσίας. Εγώ σκέφτομαι το ποινικό και το μη ποινικό δίκαιο. Μπορεί να συμμετέχει η αστυνομία στην ε, επιβολή του, ποινικού, του μη ποινικού δικαίου. Ε, Κάποιες χώρες μιλούν για αστικό δίκαιο, άλλες χώρες μιλούν για διοικητικό δίκαιο. Έχουμε λοιπόν πολύπλοκη σειρά ε, νομοθεσιών ε, στην Ευρώπη, κάτι που ε, έχει να κάνει με το τι μέτρα μπορούν να ληφθούν κατά των εγκληματιών και άλλων παραγόντων. Έχουμε ακριβώς ένα μείγμα διαφόρων ειδών νομοθετικής παρέμβασης και κάνουμε, πειραματιζόμαστε για να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα είδη νομοθεσίας. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο πειραματισμός και μας επιτρέπει να έχουμε μια ε, οπτική με πολλές αποχρώσεις. Ε, εγώ συστήνω λοιπόν ε, να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα είδη νομοθεσίας και να συνεχιστούν οι σχετικές προσπάθειες τέθηκε ερώτηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο υπάρχει πλήρης ποινικοποίηση στην πράξη των πράξεων που είναι παράνομες σύμφωνα με την οδηγία. Τα ε, στοιχεία που έχουμε μας δείχνουν ότι όχι όλες οι πράξεις που η οδηγία λέει ότι θα μπορούσαν ή πρέπει να ε, ποινικοποιηθούν ε, έχουν ποινικοποιηθεί στην πράξη ή ότι ρυθμίζονται με άλλη νομοθεσία. Υπάρχουν έγγραφα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν ότι μόνο ε, το μισό των κρατών μελών έχουν εφαρμόσει κάποιε από τις δυνατότητες που παρέχει η οδηγία. Υπάρχουν επίσης ε, κάποιες ε, αμφιβολίες σχετικά με την γνώση που αναφέρεται στην οδηγία. Σε τι βαθμό θα πρέπει όποιος έχει αποφεληθεί από θύματα ε, εμπορίας, ε, σε τι βαθμό πρέπει να γνωρίζει τις πράξεις αυτές για να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνο. Ε, σε κάποιες χώρες αυτό θεωρείται σαφής διχοτομία, δηλαδή είναι δίκαιο να, να θεωρηθεί εγκληματίας, να, να επιβληθεί ποινή σε κάποιον που γνωρίζει, ενώ σε άλλα μέρη λένε ότι εφόσον υπήρξε εκμετάλλευση αυτό είναι ε, ε, ε, κολάσιμο από μόνο του, ενώ υπάρχουν και οι ενδιάμεσες λύσεις που μιλούν για αμέλεια σε περιπτώσεις άγνοιας και υπάρχει αυτή η μέση οδός. Οι δικές μας έρευνες δείχνουν ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε το πλήρες φάσμα από την ποινικοποίηση ε, και την ε, επιβολή του νόμου ε, Υπάρχει δηλαδή μεγάλη διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κάποια αμφιβολία σχετικά με το αν το εν λόγω άτομο γνώριζε τις ενέργειες αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάγκεμαν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που τέθηκαν όσον αφορά την πολιτική ανοιχτών συνόρων. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις συνέπειες για την εμπορία ανθρώπων. Θα έπρεπε να έχουμε στοιχεία για την εμπορία πριν και μετά και δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να μπορούμε να γενικεύσουμε. Συμφωνώ ότι συχνά όταν μιλάμε για εμπορία τονίζεται η διασυνοριακή πτυχή που συνδέεται με τη μετανάστευση, αλλά όπως αναφέρθηκε, η εμπορία δεν χρειάζεται να είναι ε, καθόλου διασυνοριακή. Μπορεί μάλιστα να αφορά μια πόλη, να μην υπάρχει καμία μετακίνηση των ε, θυμάτων όπως αναφέρθηκε αυτό και πριν. Όλο αυτό συνδέεται και με το πώς μιλάμε για την ε, εμπορία ανθρώπων, ε, τι νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, ε, πώς γίνεται η αντιμετώπιση των θυμάτων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην επικεντρωθούμε αποκλειστικά σε μεταναστευτικές ροές και υπηκόους τρίτων χωρών. Είναι σημαντικό να δούμε ε, τι επικάλυψη υπάρχει ανάμεσα στην εμπορία και τις μεταναστευτικές ζωές, διότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αρκετά σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα αυτό εντός των μεταναστευτικών χωρών. Φυσικά γνωρίζουμε περιπτώσεις ε, εμπορίας ανθρώπων, δεν γνωρίζουμε όμως τα ποσοστά δεν γνωρίζουμε σε πόσες περιπτώσεις μιλάμε για εμπορία, για άλλα είδη κλιμάτων, ε, για αντικανονική μετανάστευση κλπ. Στην τελευταία μας έκθεση συμπεριλάβαμε και τη σύσταση ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσουμε στη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές και να επικεντρωθούμε και στη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα αυτών, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη δυσαναλογία ανάμεσα στα κράτη που πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, τα θύματα της εμπορίας διότι είναι σημαντικό το πρόβλημα σε περίπτωση που, κάποιος, ε, που κάποιο θύμα πάει σε χώρα που δεν έχει αρκετό δυναμικό να χειριστεί τέτοιες υποθέσεις. Όσον αφορά το θέμα των συνόρων ε, και την εγχώρια εκμετάλλευση και το αν αυτή αυξάνεται, δεν γνωρίζω αν αυξάνεται. Νομίζω όμως ότι δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα αυτό και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε το πώς εμφανίζονται τώρα περισσότερες ε, τέτοιες ε, υποθέσεις. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου και όπως αναφέρθηκε στην ε, παρουσίαση της δόκτωρος Κρούνο, θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της ασφάλειας των συνόρων. Μιλήσατε για, την, για το δυναμικό των αστυνομικών δυνάμεων και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους ε, στις κάτω χώρες. Έχουμε ομάδες της αστυνομίας που πρέπει να ασχοληθούν με διάφορα θέματα ε, και την μετανάστευση και την ε, διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν η μετανάστευση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα θα δοθεί περισσότερη προσοχή ε, στη μετανάστευση και λιγότερη στην εμπορία ανθρώπων. Και πάλι όσον αφορά την ε, εμπορία ανθρώπων βλέπουμε ότι τονίζεται περισσότερο ε, ε τονίζονται περισσότερο τα, θύματα από τη Δυτική Αφρική, δηλαδή πάλι δίνεται περισσότερη προσοχή σε αυτές τις υποθέσεις και δεν υπάρχει αρκετό δυναμικό για την εγχώρια εκμετάλλευση ανηλίκων, για παράδειγμα. Όλα έχουν να κάνουν λοιπόν με το πώς θέτουμε το πρόβλημα. Εάν ε, λοιπόν ε, βάλουμε το θέμα αυτό στο ίδιο καλάθι με τη μετανάστευση, πρέπει να βρεθεί κάποια ισορροπία και δεν είναι πάντα η σωστή ισορροπία αυτή στην οποία καταλήγουμε. Και βλέπουμε και την ε, συζήτηση στην πολιτική για την προστασία των συνόρων που συνδέεται συχνά με την ε, εμπορία ανθρώπων. Όσον αφορά την οικονομική αποζημίωση και τις οικονομικές ποινές, συχνά ε, δίδεται προσοχή στο θέμα της ανάκτησης ε, οικονομικών πόρων από τους εγκληματίες. Βλέπουμε ποινικέ υποθέσεις, έρευνες ε, για την εμπορία ανθρώπων, αλλά ήδη από την αρχή ε, των ερευνών θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, την οπτική του θύματος. Και τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία που ανακτώνται από ε, τον εγκληματία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και για οικονομική αποζημίωση του θύματος. Ε. Να μην βλέπουμε το θέμα μόνο από την πλευρά του εγκληματία, να φροντίζουμε να, ε, να τιμωρείται. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου και την οπτική του θύματος ήδη από την αρχή. Η καθηγήτρια Γόλπη ανέφερε ότι ότι είναι δυνατό ε, ε, ευρύ φάσμα μειγμάτων ε, νομοθεσίας και ποινών. Είναι σημαντικό εδώ να έχουμε κατά νου πάντα την οπτική του θύματος. Αστική ε, διαδικασία μπορεί να ε, περιορίζει πολύ το δικαίωμα των θυμάτων σε οικονομική αποζημίωση ή ακόμη και σε άδεια παραμονής. Κάποια δικαιώματα των θυμάτων εξαρτώνται από ποινικέ διαδικασίες. Ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί. Γνωρίζω ότι οι κάτω χώρες ε, έλαβαν σύσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσουν ακριβώς το θέμα της ισορροπίας στο θέμα αυτό. Δηλαδή, όταν μιλάμε για υπήκοου ε, τρίτων χωρών, ε, τα δικαιώματά τους κατά πόσο θα πρέπει να εξαρτώνται από τις ποινικέ διαδικασίε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην τελευταία ομιλήτρια και θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι. Ναι, σύντομα. Είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι η ποινική δικαιοσύνη είναι εθνική αρμοδιότητα. Η Ένωση έχει αρμοδιότητα μόνο όταν υπάρχει ένα στοιχείο διεθνές. Ε, γι' αυτό και μιλούμε για διεθνές ε, έγκλημα και μετανάστευση. Μόνο τότε υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα. Αυτό εδώ είναι το σημαντικό. Ε, για αυτό ε, το θέμα τη ε, ελέγχου της μετανάστευσης και του εγκλήματος είναι προτεραιότητα γιατί έτσι προκύπτει η αρμοδιότητα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε περισσότερα στοιχεία με το τι γίνεται με εντοπισμένα θύματα και μόλις ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία πολλές φορές κάποιοι απελάσσονται και κάποιοι και τους ε, μεταχειρίζονται ως λαθρομετανάστες. Άρα το θέμα είναι όχι τι έγινε πριν, τι γίνεται μετά. Μπορούν να μείνουν. Τα λίγα στοιχεία που έχουμε ε, καταλήγουν στο ότι θεωρούνται θύματα ε, του δηλεμπορίου μόνο κατά την ποινική διαδικασία. θύματα με την ποινική έννοια. Και, όπως είπε η Εουχένια, Αυτά γίνονται στην ε, συντηρητική πλειοψηφία των κρατών. Κυρίως εστιαζόμαστε ε, στον έλεγχο της μετανάστευσης για να καταπολεμήσουμε το δουλεμπόριο. Ναι, χρειάζεται οπτική ε, των δύο φύλων, αλλά θα πρέπει να το δούμε όσο γίνεται πιο πλατιά ή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις πολιτικές μας. Και λέει η Europol ότι εκεί που η πορνεία είναι νόμιμη ε, τότε διευκολύνονται οι εγκληματίες. Θα πρέπει να προσέξουμε με αυτά τα στοιχεία γιατί ο καθένας μπορεί να αποδείξει οτιδήποτε με στοιχεία και για να δούμε τη σχέση μεταξύ πορνείας και δουλεμπορίας είναι θέμα πολύ λεπτό. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η νομιμοποίηση της πορνείας βοηθάει το δουλεμπόριο, ούτε το ανάποδο, ούτε ότι μειώνεται το δουλεμπόριο αν ποινικοποιείται ε, ο, η συμπεριφορά του πελάτη. Τίποτα, τίποτα δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε. Ούτε προς την ούτε την άλλη κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ε, ε πάρα πολλά ζητήματα αντιφατικά ε, και δεν νομίζω ότι ωφελεί τη, τη, τη δουλειά μας τώρα να καταπολεμήσουμε δηλαδή το δουλεμπόριο με τέτοια επιχειρήματα. Δεν υπάρχει μεταξύ των δύο ζητημάτων σχέση αιτιόδου συνάφειας. Αυτά. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πόσο συμβάλλατε να έχουμε μια άποψη του τοπίου σε αυτό το περίπλοκο ζήτημα και Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε εδώ μια αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο της Αργεντινής. Είπαμε και πριν, καλώς ορίσατε. Είναι προσκεκλημένη της κυρίας Ντυπό. Επίσης, από την κάτω Σαξονία κάποιοι α, Πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της σημερινής και θα φύγουν οι προσκεκλημένες μας. Ε, ε, γεια σας. Καλώς όρισαν συνάδελφες, συνάδελφοι τέλος πάντων από την Αργεντινή. So dear, dear guests, dear ladies, where are our Argentinian uh, members, please? Ελάτε παρακαλώ οι συνάδελφοι από την Αργεντινή. So, um... Η πρόεδρος, κυρίες και κύριοι. right now, um, Συνεχίζουμε. Όπως προείπαμε, έχουμε πάρα πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά ε, τώρα να καλωσορίσουμε τους, τις προσκεκλημένες μας, βρίσκονται εδώ, εδώ και πολλή ώρα για να μας ε, ενημερώσουν ε, αυτά που ξέρουν από μέσα. Τι γίνεται στη Λατινική Αμερική γιατί πρόκειται για την προσωπική από την Αργεντινή, Σοφία Μπραμπίλα, Λορένα Ματσέν, Γκαμπριέλα Εστέβετ και Χιμένα Λόπεθ. Θα μας μιλήσουν με αυτήν την σειρά. Θα δώσουμε το λόγο, αλλά θα πρέπει να καλωσορίσουμε και τον ε, πρέσβη της χώρας ε, στο Βέλγιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εσείς καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας για αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων. Εδώ έρχονται τα νέα από την Λατινική Αμερική, μαθαίνουμε από όλες αυτές τις εκλεκτές καλεσμένες αυτά τα οποία θα πρέπει και εμείς να κάνουμε εδώ. Πρόκειται όμως για μια σπουδαία ευκαιρία ε, η οποία μας δίνεται όποτε έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Σοφία Μπραμπίλα, μπορείτε να μας κάνετε την εισήγησή σας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ. Να σας πω ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσουμε ε, σε σχέση με την νομοθεσία. Αρχίσαμε εδώ και 70 χρόνια να ψηφίζουμε και να σας πω τι γίνεται για ε, κάποια διαβήματα πολιτικά ε, και όχι μόνο τα οποία έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Εμείς οι νομοθέτες ε, μαζί με την κοινωνία κάνουμε αυτή την προσπάθεια για ισότητα ευκαιριών ανδρών γυναικών στο Κοινοβούλιο. Το 1985 κυρώσαμε ε, τα όσα προβλέπει ο ΟΗΕ για κατάργηση πάσης διάκρισης κατά γυναικών. Πάντα ήμασταν στη Λατινική Αμερική πρωτοπόροι όσον αφορά την προστασία, την ε, προώθηση της όντας των φίλων. Το 1991 εμείς και η Κωνσταντίνα ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε την πρόβλεψη του 30% κάθε ψηφοδελτίου να είναι γυναίκες. Αυτό για κάθε κοινοβούλιο ήταν παλιά 5% και μετά φτάσαμε στο 37% της συμμετοχής των γυναικών στο κοινοβούλιο. Το δε 96 με την ε, σύμβαση του ΟΕΕ Είχαμε επίσης ε, ένα νομοθέτημα για απαγόρευση πάσης βίας κατά γυναικών κάθε, κάθε μορφής βίας πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, ψυχολογικής κατά γυναικών. Ε, πρόκειται για κάποια διεθνή σύμβαση στην οποία προσχωρήσαμε, κυρώσαμε τη σύμβαση με την εθνική μας νομοθεσία και μετά φτάνουμε στο 2009. Τότε ε, θεσπίσαμε άλλο νόμο για κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το 9 είχαμε κάποια ανώτατη δικαστή που συγκρότησε το γραφείο της γυναίκας, δηλαδή μια υπηρεσία που ρύθμιζε ζητήματα ε, που αφορούν τις, τις ανισότητες. Μετά ε, το 12 είχαμε επίσης ε, τον, ε, τη, τη θέσπιση της θυπηνής των ισοβίων για γυναικοκτονία. Το 13 συνεχίσαμε το έργο μας και πέρα από την συμμετοχή στα πολιτικά, τη βία, βελτιώσαμε τις εργασιακές συνθήκες ε, όσων ασχολούνται με οικιακές εργασίες. Και έτσι ε, είπαμε ότι θα πρέπει τα οικιακά να θεωρούνται εργασία αμοιβωμένη, ε, αναγνωρισμένη και ότι πρόκειται για την πρωτοβουλία μας επομένω που την προωθήσαμε το 2013 επίσης είχαμε τη σύμβαση εργασίας για προσωπικό ε, κατοίκων για κάποιες ε, γυναίκες φτωχές που αφαιρώνουν πολύ χρόνο για τις σημαντικές οικιακές ε, εργασίες και έτσι είπαμε ότι ανοίγουμε ένα καινούριο δρόμο για την κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια είδατε ότι έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας και έχουμε επίσης κάποιους νόμους ευξημένης τυπικής ισχύω ε, για να δούμε πώς θα φτάσουμε σε αυτό το θέμα των ίσων ευκαιριών. Ε, έχουμε τις θετικές διακρίσεις βέβαια και ε, στα πολιτιστικά έχουμε παρέμβαση. Όλα αυτά είναι σημαντικά πολιτικά μέσα για να φτάσουμε στην επιθυμητή ισότητα. Το δε 17 είπαμε ότι έχουμε την ασχοληθήκαμε ακριβώ με τι ποσοστώσει εκείνε της ε, ισότητας το τριαστικό στο ψηφοδέλτιο. Σας, σας δεν είναι αυτό ζήτημα, αλλά είπαμε ότι έτσι έχουμε ε, το 50% τη ισότητα για ε, το 50% επομένως το οποίο είπαμε. 50, μισές γυναίκες, μισές άντρες για αυτούς που μπορούν να εκλεγούν και στο κογκρέσο μας από το 37 φτάσουμε το 42 και να δούμε τις επόμενες εκλογές το 2000 ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού του νόμου το 50-50 δηλαδή της εκπροσώπησης αυτά για το κογκρέσο μας και πάλι σας ε, ευχαριστούμε ε, συγγνώμη που τα είπα βιαστικά αλλά πιέζει ο χρόνος και πάλι ευχαριστούμε που καλέσατε σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η Λορένα Μαθένα έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, καλό σας απόγευμα και ευχαριστούμε που μας δώσατε την δυνατότητα και να μας ακούσετε εδώ στο Κοινοβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η ορατότητά μας ε, και γίνεται ορατή και η μάχη, ο αγώνας που δίνουμε στη Λατινική Αμερική. Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες ε, που έχουν αγωνιστεί στο στο βάθος της ιστορίας, κυρίως στην χώρα μου, έτσι ώστε εμείς να έχουμε περισσότερα δικαιώματα, περισσότερες ευκαιρίες και να καταφέρουμε αυτό που έλεγε η Σοφία προηγουμένως και νομίζω ότι όλοι, ε, όλοι συμφωνούμε με αυτό, δηλαδή ότι ε, όλοι οι πολιτικοί ηγέτες ε, ε, γυναίκες πολιτικοί, βουλευτές, ε, αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να γίνει δεχτή η διαφορετικότητα, γιατί αυτή η διαφορετικότητα θα μας ε, κάνει καλύτερες κοινωνίες, θα βελτιώσει τις κοινωνίες μας. Εμείς βλέπουμε την Ευρώπη σαν ένα παράδειγμα από την Λετινική Αμερική και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σε όλα αυτά τα θέμα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια γυναίκα η οποία κατάφερε να αγωνίζει όταν ε, ο αγώνας αυτό ήταν ε, αδύνατος. Ε, η Φιωρεντίνα Γκόμες Μιράντα, πολιτική γυναίκα της, από την Αργεντινή, που προώθησε πολύ τα δικαιώματα των γυναικών για θέματα ας πούμε των διαζυγίων, την δυνατότητα διατήρησης δικαιωμάτων μέσω των γαμικών συμβολέων, καθώς επίσης ε, την δυνατότητα της ε, ε, διακοπής κοίησης. Όταν τα έκανε όλα αυτά η Φιωρεντίνα ήταν πραγματικά σαν να βρομόλογα βρωμόλογα το να μιλάς για τέτοια πράγματα στην Αργεντινή και όμως άνοιξε την κουβέντα στην Αργεντινή. Ε, ΑΚΕ οδήγησε στην Αργεντινή στη συζήτηση για το δικαίωμα που έχουμε ε, ε, πάνω στα, στα σώματά μας και επίσης και για άλλα θέματα όπως ας πούμε το μισολογικό φάσμα, χάσμα συγγνώμη, που, στο οποίο αναφέρθηκε η Σοφία προηγουμένως. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου γίνεται αυτή η συζήτηση που μας απέδειξε ότι όταν μία γυναίκα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου υφίσταται μία συμπεριφορά η οποία ε, είναι βία, η οποία ε, παραβιάζει τα δικαιώματά της, τότε αυτό δεν αφορά μία συγκεκριμένη γυναίκα σε μία συγκεκριμένη χώρα. Ε, θα πρέπει να δούμε σαν να είμαστε πραγματικά ε, ε, ε, με ενσυναίσθηση απέναντι να στεκόμαστε σε αυτές τις γυναίκες, σαν να είμαστε αδερφές και επομένως πρόκειται και για ένα θέμα ή για θέματα τα οποία θα πρέπει εγκάρσια να απασχολούν όλα τα πολιτικά κόμματα. Εμείς γυναίκες πολιτικοί σε συνεργασία με κοινωνικές οργανώσεις καταφέραμε να επιτύχουμε ένα υψηλό βαθμό ηθικής δεοντολογίας θα ήθελα να πω. Και ε, ε, τελικά ε, είχαμε μια συζήτηση πολύ υψηλού επίπεδου που μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε τις γυναίκες από διαφορετικό πρίσμα και λαμβάνοντας υπόψη άλλες παραμέτρους, εστιάζοντας στο πώς είμαστε και στο πώς μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να έχουμε καλύτερες, περισσότερες ευκαιρίες στο μέλλον. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, ωστόσο θα ήθελα ε, να προβληματιστούμε, να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε το εξής. Αυτός ο ε, αιώνας είναι ο αιώνας των γυναικών. ιδιαίτερωση εις την ε, ε, Αργεντινή από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας του 1983 μέχρι τώρα μας έχει... Έχουμε πολλές ε, ουσιαστικές βελτιώσεις, νομοθετικές, θεσμικές ε, στην καθημερινή ζωή. Ο αγώνας θα συνεχίσει ε, και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα που πρέπει να είναι ένας αγώνας που θα ξεπερνάει τα σύνορα, που θα ξεπερνάει τις πολιτικές ιδεολογίες και τα πολιτικά ε, σύνορα και θα πρέπει να αφήνει πίσω της ε, η διαδικασία αυτή την ε, υποκρισία και να μην λησμονεί και την διάσταση της δημόσιας υγείας, γιατί η δυνατότητα νόμιμης διακοπής κοίησης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε πια γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους σε παράνομες ε, διακοπές ε, κοίησης. Ε, θέλουμε να αποφύγουμε καταστάσεις όπου οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν αρκετά χρήματα ήταν υποχρεωμένες να το κάνουν παράνομα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καπριέλα Εστεβές, παρακαλώ. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Λιδία, την Μόνικα για την ε, πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας τιμή να έρθουμε εδώ να σας πούμε την εθνική μας ε, εμπειρία να είμαστε εδώ σε ένα τέτοιο κοινοβούλιο. Για να δούμε λίγο περισσότερο ε, τι ακριβώς σημαίνουν όλα όσα έχουν γίνει για το γυναικείο κίνημα. Το ότι είμαστε εμείς εδώ και μιλούμε έχει σχέση με τις συνέπειες των όσων έγιναν στην χώρα μας. Έχουμε 30 χρόνια που γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, γίνεται όλη αυτή η συσπήρωση των γυναικών ε, όσον αφορά ε, τις ε, αμβλώσεις στο θεματολόγιο και τα άλλα θέματα όλα αυτά ε, το, το, για το πώς θα συγκρομινοποιηθούν, θα υλοποιηθούν τα δικαιώματά μας και θα εκπροσωπηθούμε κοινοβουλευτικά. Ε, αυτό είναι παλαιό θέμα, επομένως αλλά αναδύθηκε στη δημόσια ε, ζωή πρώτα-πρώτα με αυτό το κίνημα. Το κίνημα των γυναικών που έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις αλλά ξεκίνησε και στην Αργεντινή με την καταπολέμηση της γυναικοκτονίας. Και ακριβώς ε, έχουμε κάποιες εθνικές στατιστικές και διεθνείς σε σχέση με αυτά τα θύματα, αυτές τις γυναίκες κάθε 28 ώρες ότι πεθαίνει μία γυναίκα στη χώρα μας και αρχές της χρονιάς είχαμε μία γυναίκα ανά 22 ώρες μία γυναίκα θύμα γυναικοκτονίας και ξεκίνησε στο, στο πεζοδρόμιο το, το, το κίνημα από το 2015 θεωρήθηκε ότι είναι κατεπήγον θέμα κάτι να γίνει για τη βία κατά των γυναικών, διατέθηκαν για πρόληψη και δημοσίου πόροι, ευαισθητοποίηση ε, και η συζήτηση άναψε λοιπόν και όλο ένα επομένως και εξετάζεται το ότι έχουμε αυτή τη βία αυτή τη βία που είναι κάτι σαν πολιτιστικό φαινόμενο και κοστίζει ζωές κάθε μέρα. Ε, Οπότε λοιπόν χτίστηκε αυτό το κίνημα και αυτά μπήκαν ε, στην δημόσια προβληματική όλα τα ζητήματα σχετικά με την βία κατά των γυναικών. Και ήταν και το θέμα των αμβλώσεων, το οποίο ήταν από τα πιο σημαντικά. Γιατί να, η μια τρομερή βία κατά του σώματός μας. Ε, όλα αυτά παράνομα και όλα αυτά έχουν ευξημένη συμβολική σημασία για την βία κατά των γυναικών, τόσων γυναικών που πέρναγαν από τόσες, ε, τόση παρανομία ε, και ε, επειδή ήταν τόσο παράνομες, ήταν παράνομες οι αμβλώσεις υφίστανται ότι υφίστανται οι γυναίκες ε, δεν υπήρχε νομοθεσία ή δεν είχαν χρήματα να κάνουν νόμιμη άμβλωση οπότε τελικά πρόκειται περί βίας βίας από πλευράς του κράτους εις βάρος του γυναικείου σώματος και έτσι λοιπόν φούσκωσε αυτό το κίνημα συσπήρωση ε, αφορούσε τις πιο νέες ε, γυναίκες. Βλέπω ότι έχω εδώ πολλές τέτοιες γυναίκες και στην Αργεντινή. Ε, οι πιο μεγάλες πρωταγωνίστες ήταν οι νέες. Μιλούμε για γυναίκες από τα 13, σχεδόν παιδιά, που κατέβηκαν στο πεζοδρόμιο για να μπορέσουν να έχουν την διαχείριση, την αυτοδιαχείριση του κορμιού τους τελικά όσον αφορά ε, το να μπορούν να πάνε δωρεάν και με σιγουριά να κάνουν την άμβλωσή τους σε κέντρα θεσμικά. Ε, και στη συνέχεια ε, όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά πολιτικά και όλα αυτά μπήκαν και στο κοινοβουλευτικό θεματολόγιο και επί δύο προέδρων της Δημοκρατίας από δύο διαφορετικές πολιτικές πτέρυγες αυτή ε, έβραν λοιπόν στο θεματολόγιο την ε, άμβλωση και συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο. Οπότε αυτή η δύναμη του γυναικείου κινήματος που είχε τέτοιες διαστάσεις ε, όλα αυτά πήγανε στο Κοινοβούλιο και είχαμε φεμινίστριες βουλευτίνες που τώρα έχουμε σηκώσει αυτή την σημαία για να δουλέψουμε το θέμα στο Κοινοβούλιο, να υπάρχει οριζόντιος χαρακτήρας, διακομματικός, ε, γυναίκες κάθε ηλικίας, ακριβώς όπως τα είπε η προλαλήσασα, ε, να συζητήσουμε σαν αδελφές, ε, ισό με ισότητα και με συμμετοχή από κάθε κατεύθυνση, με κάθε είδους επιχειρήματα υπέρ και κατά, να το φτάσουμε το θέμα στο τέρμα του για να πετύχουμε αυτήν την ιστορική παραχώρηση ή κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Να, το πετύχαμε αυτό στο Κοινοβούλιο. Επίσης είχαμε κάποια προβλήματα και στην, ε, ε, στη Γερουσία και τελικά όμως ε, επειδή υπήρχε πρόβλημα στη Γερουσία κατέβηκαν στο δρόμο δύο εκατομμύρια γυναίκες από παντού, από κάθε γωνιά και ε, τομέα της κοινωνίας ούτω ώστε να λάβει σάργα και οστά το δικαίωμά μας αυτό είπαμε για την εκπροσώπησή μας την κοινοβουλευτική εσείς αυτά τα ξέρετε γιατί το είχατε αυτό δεδομένο. Ε, ε, με εμά όμως και σε εμά έτσι έγινε. Όλες, όλες οι γυναίκες που δυσάγγιζε αυτό το πρόβλημα ήταν ένα κοινωνικό αίτημα. Ήταν λοιπόν μια στρατηγική συμμαχία. Αυτό το πετύχαμε ως κίνημα γυναικείο. Είπαμε διακομματικό, γυναίκες κάθε ηλικίας, αλλά έτσι κερδίσαμε και τους ε, χώρους ε, της κοινωνίας που ασχολούνται με τη διαφορετικότητα, την σεξουαλική. Ε, όλοι όλοι είχαν το φεμινιστικό στοιχείο. Οπότε έτσι προχωρήσαμε και σε νόμους που προστατεύουν τους διεμφυλικούς σε σχέση με την εργασία για να έχουμε ρυθμίσεις ε, συνεκτικές, οριζόντιες και αυτό κέρδισε όλους τους πολιτικούς χώρους. Προωθήσαμε ένα σωρό νομοσχέδια με αδελφικό πνεύμα. Για όλα αυτά τα δικαιώματα που πρέπει να αναγνωριστούν, τα δικαιώματα αυτά να ενσωματωθούν σε νόμο να έχουμε μια πιο δημοκρατική κοινωνία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κινάρα Λοπές. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να κλείσω λίγο αυτά που είπαν οι συναδέλφισές μου. Όλες βεβαίως είμαστε αγωνίστριες ε, στρατευμένες στο θέμα το, στα γυναικεία ζητήματα, στην, στο θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ιδέα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό ακριβώς, ε, παρότι προερχόμαστε από διαφορετικά κόμματα, διαφορετικά ε, του ιδεολογικού φάσματος. Παρ' όλα αυτά είμαστε αδερφές όσον αφορά αυτό, αυτά τα θέματα. Ε, ξέρετε ότι η Αργεντινή ε, είχε να αντιμετωπίσει μία από τις πιο σκληρές δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής που απήγαγε ε, μικρά παιδιά και λοιπά και που από το 83 ξεκίνησαν οι διαδικασίες που έγιναν γνωστές ως οι γυναίκες και οι γιαγιάδες της πλατείας του Μαΐου ήταν ιστορικές οι στιγμές ε, και οι γυναίκες εμείς κατεβήκαμε στους δρόμους ε, ε, και ήταν τότε με την υπόθεση Κουτράλκο και άλλαξε ο τρόπος ε, με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα φεμινιστικά θέματα, τα ζητήματα των γυναικών ε, χωρίς ε, ιδεολογικούς περιορισμούς, χωρίς σύνορα κτλ. Ξεκινήσαμε τότε ακριβώς να συζητούμε για θέματα που αφορούν τις γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό πρότυπο, το κοινωνικό πρότυπο της Αργεντινής, το κοινωνικό πρότυπο της ενσωμάτωσης μετά από ε, χρόνια ε, πολέμου και ε, βίαιης αντιμετώπισης και τότε έπρεπε να δημιουργήσουμε πολιτικές, κοινωνικές πολιτικές, να ξεφύγουμε από πολιτικούς κύκλους που εν τέλει άφηναν την χώρα με πολύ αυξημένο χρέος. Στην Αργεντινή είχαμε την δυνατότητα να έχουμε ένα Υπουργείο Ε, γυναικών και ε, κοινωνικής ανάπτυξης που δημιούργησε ο τελευταίος ε, πρόεδρος Φερνάντες. Αρχίσαμε να συζητούμε για την πολιτική με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή ξεπεράσαμε αυτήν την, αυτόν τον κατακαιρματισμό της πολιτικής, τα κουτάκια τα οποία αποτελούν την πολιτική και είπαμε ότι θα πρέπει με τρόπο πιο συνολικό να προωθεί βοηθήσουμε την ε, πολιτική και τη χώρα. Ε, επίσης, το τέταρτο πράσινο κύμα που περιλαμβάνει το φεμινιστικό κύμα είναι αυτό ε, το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη του φεμινισμού μέσα στις δομές ε, του, τις εκτελεστικές δομές ε, του κράτους που έδωσε την δυνατότητα να αλλάξουμε την πολιτική σκέψη, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονταν οι προϋπολογισμοί στην Αργεντινή. Είχαμε λοιπόν την δημιουργία αυτού του συγκεκριμένου Υπουργείου ε, που απέκτησε ε, ειδική εξουσία που σχετίζεται ε, και με το ξεπέρασμα των παλαιών κουρασμένων πολιτικών του κατακαιρματισμού. Μια ε, λογική λοιπόν που αλλάζει σε όλα τα Υπουργεία που βασίζεται βεβαίως η αλλαγή αυτή σε υπαλλήλους, ε, γυναίκες υπαλλήλους ε, που έχουν καταρτιστεί η Ελένη Καέλα είναι ε, αποτέλεσμα μιας ε, πολύ σκληρής ε, διαδικασίας που ξεκίνησε από την γυναικοκτονία της Μικαέλα Θέρα. Ο πατέρας της με τον οποίο έχω και προσωπικές σχέσεις ο, επέμεινε έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει, να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες αυτής της ε, γυναικοκτονίας. Ήταν μια νέα γυναίκα ε, η οποία σπούδαζε γυμνάστρια, ε, ήταν φοιτήτρια φυσικής αγωγής και που έχασε την ζωή της. Και μετά δημιουργήθηκε ένας νόμος που έδωσε την δυνατότητα της διάστασης φίλου σε φίλου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους τομείς. Ε, ε, άρχισε λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την πατριαρχία, με το φίλο, ε, την σεξουαλική παρενόχληση, την ιδιαίτερη βία λόγω του φύλου κλπ. Και δόθηκε ακριβώς η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε στη η διάσταση του φύλου μέσα από την ίδια τη δυναμική αυτή τη διάσταση. Και ε, γι' αυτό ακριβώ ε, εμεί ε, ζητούμε στα ίδια τα πλαίσια αυτή τη συζήτηση ε, την νομιμοποίηση της ε, γιατί θα αποτελέσει, αν θέλετε, και το επιστέγασμα μιας χρόνιας διεκδίκηση. Εμείς θέλουμε μία φεμινιστική λογική ε, η οποία δίνει την δυνατότητα η διάσταση φύλου να παίξει κεντρικό ρόλο σε όλες τις ε, λαϊκές ε, πολιτικές, κυρίως δε για να ληφθούν υπόψη γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, βία, οικονομική βία κλπ στις 45-50 μέρες της δημιουργίας ε, του Υπουργείου που ανέφερα προηγουμένως είχαμε την ε, δυνατότητα να δούμε να θεσπίζεται ένα εθνικό σχέδιο το οποίο λαμβάνει υπόψη ε, Ε, να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που ε, ε, δαπανούμε για να προστατέψουμε, να προσέξουμε, να ασχοληθούμε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και εμείς θέλουμε αυτού του είδους ε, η εργασία ε, να μπει σε ένα πλαίσιο ε, πιο καλά ρυθμισμένο, σε ένα επίσημο σχέδιο, γιατί έχουμε 30% ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και το 50% τουλάχιστον αυτών των ανθρώπων είναι γυναίκες. Ε, η φτώχεια λοιπόν έχει γυναικείο πρόσωπο στην Αργεντινή και επομένως θα πρέπει να δοθούν δυνατότητες στις γυναίκες μέσα από ένα σύστημα ενδεχομένως όπου θα αμείβεται αυτή ε, η ε, φροντίδα που δίνουν σε άλλους ανθρώπους. Επίσης να δούμε τις γυναίκες οι οποίες δουλεύουν σαν οικιακές βοηθοί γιατί πρόκειται για γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτωχοποίησης. Ε, πολλές πρωτοβουλίες λοιπόν λαμβάνονται και γι' αυτό στρεφόμαστε και προς ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς τις ε, ισπανόφωνες βουλευτίνες που μας έδωσαν την δυνατότητα να έρθουμε εδώ. Ε, υπάρχουν πολλά ζητήματα που είναι ανοιχτά, αλλά για μας ε, η εθελούσια διακοπή κοίησης, ε, η άμβλωση με νόμιμο, σε εθελοντική βάση και με νόμιμο τρόπο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες έχουν ζήσει πολλά, οι οποίες έχουν περάσει από φτώχεια, από βασανιστήρια, από την αδυναμία να ασκήσουν τα πολιτιακά τους δικαιώματα ε, και επομένως ε, ζητάμε για όλες αυτές τις γυναίκες την προστασία του κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ευρία επισκόπηση της κατάστασης που μας δώσατε. Υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων η Σέρβος Ραφαέλα και μετά η Μόνικα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Χαίρομαι γιατί είμαι και πρόεδρος του Φόρουμ των Γυναικών στην Eurolat και θα έρθω σε επαφή με μαζί σας να μιλήσουμε και αύριο. Αλλά είναι καλή ευκαιρία που σας έχω σήμερα εδώ να σας πω ξεκάθαρα ότι βεβαίως εδώ είμαστε... Ε, ε Είμαστε γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας υποστηρίζουμε στις προσπάθειές σας. σε θέματα παρενόχλησης γυναικών, εκφοβισμό γυναικών, ε, κυρίως στην πολιτική. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε κάτι συγκεκριμένο που σκέφτεστε να κάνετε έτσι ώστε να ε, δείξετε ότι ο εκφοβισμός και η ε, παρενόχληση των γυναικών είναι, πρέπει να σταματήσει κυρίως στην πολιτική αλλά όχι μόνο. Και δεύτερο, Πρόσφατα ήμουν στον Παναμά με την αντιπροσωπεία Eurolat και έκατε σαφές ότι υπάρχουν και προκλήσεις ας πούμε για τις ε, αφρολατίνες γυναίκες, για τις ε, γυναίκες ε, ε, τις, αυτόχθονες. Άρα να ρωτήσω τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να βελτιωθεί η θέση των ε, ειδικών αυτών ομάδων ε, των γυναικών στην χώρα σας και στη Λατινική Αμερική γενικά. And then Maria Manuel. Μαρία Μανουέλ. I just, I make one after the other. Όλες με τη σειρά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εννοείται να ευχαριστήσουμε και τις προσκεκλημένες, τις τέσσερις συναδέλφους από το Αργεντίνικο Κογκρέσο. Μπράβο για το διακομματικό χαρακτήρα της αντιπροσωπείας, γιατί η καθεμία σας προέρχεται από διαφορετικό κόμμα, αλλά είστε συσπηρωμένες. Στο όνομα των δικαιωμάτων της γυναίκας. Και ευχαριστούμε και το, το επιτελείο της πρεσβείας της ε, χώρας και όλους όσους ήρθαν εδώ και βοήθησαν. Σένα ευχαριστούμε, Πρόεδρε, που το έκανες αυτό και που δεν όλα αυτή, αυτό το, τον αγώνα για κάτι τόσο σημαντικό για το γυναικείο σώμα. Θέλω να σας ρωτήσω, βέβαια είναι ξεκάθαρο αυτό που μας είπατε για το κοινωνικό κίνημα που γεννήθηκε στην Αργεντινή, να σας πω Κάτι που πάντα λέει η Γκαμπριέλα Σερούτη, διάσημη ε, κοινοβουλευτικός, ε, ότι προερχόμαστε από τους Λευκούς και στρεφόμαστε προς τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας σε κάθε γωνία της χώρας. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι προβλέπετε, τι επόμενα βήματα θα κάνετε. Θα δουλέψει το κοινοβούλιο σας τώρα ε, μέχρι τον επόμενο μήνα, πότε θα έχετε διακοπές, ε, τι θα κάνετε, θα εξουπίσετε το χρόνο σας. Τι, μπορεί, τι νομίζετε ότι μπορούμε εμείς κάτι να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε στον αγώνα σας. Ε, thank you, Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να σας τα πω στα ισπανικά. Πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσουμε Μόνικα και για όλες τις προσπάθειες τώρα που έχετε αυτό το μικρό διάλειμμα για όλη σας την προσπάθεια μπράβο και στην Εβελίν Ρέγνερ μόλις προτείναμε να γίνει η πρόσκληση ευθύς αμέσως μας βοήθησε και τη Μόνικα και εμένα μπράβο Εβελίν ευχαριστούμε ξεπέρασες την παραδοσιακή μας γραφειοκρατία. Πολύ σημαντικές αυτές οι συναντήσεις. Να έχουμε ανταλλαγές απόψεων, να δικτυωθούμε όσον αφορά τον αγώνα για ισότητα, αυτονομία, αξιοπρέπεια για το σώμα της γυναίκας που είναι αγώνας παγκόσμιου χαρακτήρα. Υπάρχουν οι ιδιοτυπίες, οι εθνικές, η καθεμία βρίσκεται αλλού. Είναι θέμα φιλής, κοινωνικής τάξης, θέμα γεωγραφικό. Είναι αγώνας για να έχουμε την εξουσία πάνω στο σώμα μας. Αλλού παλεύουμε για την άμβλωση, αλλού το να μην ε, είναι νόμιμη υποκατάστατη μητέρα αλλού δίνεται αγώνα για τις γυναίκες με αναπηρία, ε, στις Αμερικανικές φυλακές γίνεται στήρωση αναγκαστική, αλλού είναι τόσο φτωχές γυναίκες, δεν μπορούν να γίνουν μάνες, αλλού υποχρεούνται να γίνουν μάνες γιατί αλλιώς ε, έχουν το κοινωνικό στίγμα. Οπότε όλα αυτά είναι κομμάτι του ίδιου αγώνα. Αυτό να κάτσουμε να δούμε. Τις διαφορετικές πτυχές του αγώνα μας σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Αυτά να συνειδητοποιήσουμε. Το χρειαζόμαστε. Η συνειδητοποίηση είναι απαραίτητη. και ε, βέβαια. Και εμείς αυτά τα πιστεύουμε, αλλά και αυτούς που δεν πιστεύουν θα πρέπει να τους πείσουμε. Αλλά για την συνειδητοποίηση τι χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να προωθήσουμε το φεμινιστικό κίνημα, όπως τα είπε και η Μόνικα, ότι εσείς, εσείς είσαστε παράδειγμα προς μίμηση για το γυναικείο κίνημα, τα δικαιώματα των γυναικών, για τη δημοκρατία. Η Αργεντινή είναι επίσης παράδειγμα του πόσο οι γυναίκες παλεύουν για την δημοκρατία. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι θρεμοσβήνει η φλόγα της δημοκρατίας σε πολλά μέρη του κόσμου. Γιατί έχουμε καταπίεση της γυναίκας, έχουμε κίνημα αντιφεμινιστικό. Άρα είναι σημαντικές οι προσπάθειες του δημοκρατικού κινήματος και είναι κρίσιμες οι ώρες να ενωθούμε, να συζητούμε, να δικτυωθούμε. Για ισότητα, αξιοπρέπεια για το σώμα μας, για την αυτονομία μας. Είναι αγώνα στην πρώτη γραμμή. Για τη δημοκρατία. Άρα, να συνθούμε και να ξανασυναντηθούμε. Και όπως είπε η Μόνικα, πέστε μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Τι να κάνουμε εμείς. Uh, Ευχαριστώ, Μαρία Μανουέλ. Και μετά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα τα πω στα πορτογαλικά. Θα αλλάξω γλώσσα. Είμαι συντονίστρια για την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών όσον αφορά τη Eurolat και είμαι και μέλος της παρούσας επιτροπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τους αγώνες που κάνετε στις δικές σας χώρες, ε, για τους οποίους μας μιλήσατε εδώ σήμερα. Είμαι βέβαιη ότι έχουμε ακούσει μόνο λίγες πτυχές ε, της δουλειά σας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο στους αγώνες αυτούς. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε τον ε, ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Είναι κάτι που ε, συμβαίνει και, στη και στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και δεν, θα πρέπει να έχει εξαλειφθεί από όλα τα σημεία του κόσμου. Ασχολούμαστε και με άλλα θέματα. Στη χώρα μου ε, είχαμε δύο δημοψηφίσματα για να νομιμοποιηθούν οι αμβλώσεις. Ε, την πρώτη φορά χάσαμε και έπρεπε να ξαναθέσουμε το θέμα για να αποποινικοποιηθούν οι αμβλώσεις. Μπορούμε να είμαστε υπέρ ή κατά, αλλά δεν επιτρέπεται να αποτελεί έγκλημα τη στιγμή που ε, πεθαίνουν ε, γυναίκες σε σκοτεινά κλιμακοστάσια επειδή δεν κάνουν ε, σωστή άμβλωση. Κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο στο σημερινό κόσμο. Το βλέπουμε στην Ευρώπη σήμερα. Βλέπουμε να πρέπει να αγωνιζόμαστε για δικαιώματα που θεωρούσαμε δεδομένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε συνεχώς, να επαγρυπνούμε, διότι δεχόμαστε συνεχώς ε, πιέσεις. Πρέπει να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να αποφύγουμε τις ανισότητες. Ε, μπορεί να μην είναι τα πιο επίκαιρα θέματα στη δημόσια συζήτηση, αλλά ε, μπορεί να είναι χρήσιμο να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Επίσης, δεν βλέπουμε πολλές γυναίκες ε, στην τεχνολογία και αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα στο μέλλον, ε, διότι είναι συχνά οι καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και θα είναι αποφασιστική σημασία στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ε, εξαρτηστούμε με το θέμα αυτό σήμερα για να μην χρειαστεί να αγωνιστούμε για αυτό στο μέλλον. Όσον αφορά την Eurolat, ήμουνα τον Δεκέμβριο στον Παναπά και πρέπει να πω ότι αυτό ήταν το καλύτερο τμήμα όλης της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης. Ακούσαμε τα προβλήματα των Λατινοαμερικανών γυναικών. Ανταλλάξαμε εμπειρίες και ήταν πολύ ενδιαφέρον τμήμα της όλης συζήτησης και θα ήθελα να συνεχίσουμε τις εργασίες αυτές ώστε κατά την επόμενη Eurolat, ε, κατά την επόμενη διακοινοβουλευτική συνέλευση Eurolat ε, στο Σανταφέ στην Αργεντινή, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω σε κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν σήμερα. Μπορείτε να βασίζεστε στη δική μας αλληλεγγύη. Όλα αυτά τα θέματα, ακόμα σε περιπτώσεις όπου μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον αγώνα τουλάχιστον σε κάποια κράτη-μέλη, ε, μπορεί συνεχώς να ξανατίθενται στο θεματολόγιο και να απαιτούν νέους αγώνες. Ευχαριστώ, Ηλιά. Ε, Καλό απόγευμα σε όλους. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και που κάνετε ακουστή τη φωνή σας και γνωστό τον αγώνα σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας αυτός ε, και όταν κερδίζει μια χώρα τον αγώνα αυτό, ένα σημείο τον αγώνα αυτό, ε, τελικά με την, με την ιδέα αυτή του φαινόμενου της πεταλούδας και άλλες χώρες επηρεάζονται. Ε, μέσω της Eurolat ε, πριν εδώ και χρόνια ε, οργανώνουμε στα πλαίσια του Eurolat ημέρες, ημερίδες μάλλον για την ε, γυναικοκτονία. Σε λίγο καιρό θα οργανωθούν ε, αυτές οι ημερίδες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ε, και να αντιμετωπίσουμε είναι την, τη μορφή βίας στην Αργεντινή, στο Μεξικό, σε όλες τις χώρες ε, το θέμα ε, επίσης ε, της πολιτικοδικαστικής βίας, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάρτιση που είναι τόσο σημαντική στην αστυνομία, στον δικαστικό κλάδο, πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι καινοτομίες στις ομάδες που θα πρέπει να είναι θεραπενίδες και αρρωγή οδηγεί μάλλον στον αγώνα μας. Εμείς ε, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε επαφές μεταξύ μας ε, και αν ε, έχετε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, κάποιο σημείο που θέλετε να συμπεριληφθεί σε αυτή τη συζήτηση για τις γυναικοκτονίες και την βία της αστυνομίας και του δικαστικού, παρακαλώ να μας δώσετε. Η ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συντρόφισσες που μας ε, ε, κάλεσαν και βεβαίως να ευχαριστήσω την Ευελίν ε, που πάντα είναι διαθέσιμη. Εγώ Έμαθα πολλά από την εμπειρία που είχα στην ε, Αργεντινή. Πολύ μεγάλος παραλληλισμός μπορεί να υπάρξει ανάμεσα ε, στον ε, αγώνα που δίνουν οι γυναίκες στην Αργεντινή και στην Ισπανία. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις οι τωρινές και στην Ισπανία και στην Αργεντινή ε, με επικεφαλής ε, την Μοντέρο στην Ισπανία. Ε, έχουμε λοιπόν λέω τα Υπουργεία τα οποία ασχολούνται με τα θέματα αυτά, με επικεφαλής την Μοντέρο στην Ισπανία και αντιστοίχως και στην Αργεντινή και πραγματικά με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προωθήσουμε και όλα τα φεμινιστικά θέματα και βεβαίως να να ζητήσουμε και από την Ρούτη και την Οφέλια Φερνάντες ε, να έρθουν κάποια στιγμή ε, και νομίζω ότι ήταν και η πιο νέα βουλευτής ε, της Λατινικής Αμερικής. Αυτό που ρώτησε η συνάδελφος Σαμίρα που είναι ενδιαφέρον να μας πείτε τι γίνεται με την πολυεθνικότητα Ε, ο αγώνας της Μιγιάν, πώς εστιάσατε ε, στα θέματα αυτά από πλευράς θεσμικών οργάνων. Γιατί, κοιτάξτε, εγώ είμαι φεμινίστρια, είμαι στρατευμένη, τώρα είμαι ε, Ευρωβουλευτής αλλά ήμουν και καθηγητής για για θέματα φύλου κλπ. Αυτό το θέμα της πολυεθνικότητας μπορεί να αποτελέσει σημείο τριβής και έντασης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε πώς το αντιμετωπίσατε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Το έλεγε και η συνάδελφος Σαμίρα, ε, σας ε, υποστηρίζουμε αναμφίβολα αλλά έχουμε κάποιες δυσκολίες να μιλήσουμε για ε, σεξουαλικά δικαιώματα, δικαιώματα αναπαραγωγής και να βάλουμε, να εντάξουμε τις αναφορές αυτές στα κείμενα. Το Κοινοβούλιο είναι σαφές όσον αφορά τα θέματα αυτά, αλλά ε, το Συμβούλιο ε, ανθίσταται πολλές φορές κυρίως μέσω της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και στην Ισπανία και θα τελειώσω με αυτό. Έχουμε ένα πρόβλημα γιατί και σε, σε σχέση με αυτό που έλεγε και η συντρόφισσα προηγουμένω, το θέμα τη ε, άμβλωσης έχει αντιμετωπιστεί αρκετά σωστά. Ωστόσο, σε μία προσφυγή ε, στο δικαστήριο, στο ανώτατο δικαστήριο υπάρχει το όριο των 14 ε, εβδομάδων. Έχουμε ακόμα και το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ε, σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία και αυτό το θέμα της σύμφωνης γνώμης των γονέων. Ε, αυτά όλα είναι λίγο αγκάθια τα οποία μας προβληματίζουν. over questions and comments. Uh, Ακούσατε λοιπόν ε, ερωτήσεις ε, και παρατηρήσεις. Θα ήθελα και εγώ να θέσω μια ερώτηση. Σε εποχές που σε πολλές χώρες αντιμετωπίζουμε μια εθνική αντίδραση. Είναι πολύ σημαντικό να είστε εδώ και να έχουμε τέτοιες ανταλλαγές ε, σχετικά με τα θέματα όπου έχουμε πρόοδο, διότι οι αντιδραστικοί ε, έτσι θέτουν το πρόβλημα. Εάν λοιπόν εμείς ε, παρουσιάσουμε τις δικές μας θετικές ιστορίες, μπορούμε να πούμε ορίστε. Έχουμε εξαιρετικές γυναίκες από την Αργεντινή που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιχείρημα για όλη την πολιτική μας δουλειά. Από την άλλη είναι εξαιρετικό το ότι έχουμε τέτοιες ανταλλαγές απόψεων και θα ήθελα να σας πω ότι... Το πρωί είχαμε την, ε, ε, την σύσταση του δικτύου ε, για τη συμπερίληψη της διάστασης ε, των δύο φύλων ε, σε όλες τις πολιτικές. Θα ήθελα να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και για τις τεχνικές στοιχές. Πώς λειτουργεί η ενσωμάτωση της διάστασης των δύο φύλων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς έχουμε αρμόδιους εισηγητές σε όλες τις επιτροπές που τονίζουν θέματα όπως είναι η σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και ενσωμάτωση της διάστασης των δύο φύλων ε, στον προϋπολογισμό, για να γνωρίζουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα. Ε, είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο να έχουμε ανταλλαγές ε, απόψεων για τα θέματα αυτά και είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στις μελλοντικέ μας εργασίες. Ως Ευρωβουλευτές βλέπουμε ότι σε κάθε επιτροπή είναι διαφορετικά τα πράγματα και πάντα μπορούμε να παίρνουμε ιδέες και να έχουμε ανταλλαγές απόψεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν προς εσάς. Και πέρα από το gender mainstreaming, την ενσωμάτωση της διάστασης των δύο φύλων, ε, στο ε, μέλλον ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Στη Eurolat, που είναι κάτι πρακτικό, είναι κάτι υπάρχον. Και σε επίπεδο ΟΗΕ, τι μπορούμε να κάνουμε. Οι γυναίκες θα πρέπει να είναι ενωμένες από όπου και να προέρχονται. Οι γυναίκες ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική και στην ε, Ευρώπη ε, μοιραζόμαστε ε, την ίδια κουλτούρα. Θα ήταν εξαιρετικό λοιπόν εάν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και σε τεχνικό επίπεδο. Και σας ξαναδίνω το λόγο με τη σειρά που ξεκινήσαμε. Πρώτα η κυρία Μπαμπίλα. Σοφία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ συγκεκριμένα θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση ακριβώς. Πρόκειται για την πολιτική βία, για είναι κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει αρκετά, διότι ε, στο κόμμα μου, στη χώρα μου είμαι εγώ η αρμόδια για το θέμα αυτό, το, το γυναικείο θέμα και όσον αφορά λοιπόν την ε, συμμετοχή μας στα πολιτικά. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ επίκυρο το ζήτημα και το συζητάμε συνέχεια την πολιτική βία. Και σήμερα στο πάνελ είδαμε το ότι πρέπει να αρθούν αυτοί οι φραγμοί. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ε, αμφιβολία ότι εμείς μπορούμε, είμαστε έτοιμες για αποφάσεις, για ευθύνες και θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό νομίζω ότι το κοινό μας θέμα είναι το πώς αυτά θα τα βάλουμε κατά μέρος, πώς ε, θα σταματήσουμε και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα το φράγμα κατά των γυναικών. Ε, και οπότε είπαμε για το νομοθεσία, για την προστασία των γυναικών από τη βία και να δούμε πώς θα ξεριζώσουμε την πολιτική βία. Τα είπαμε στο κόμμα και είπαμε ότι συνέχεια, συνέχεια ανακύπτουν τα ζητήματα ε, θα πρέπει να δοθεί απάντηση από όλο το πολιτικό φάσμα. Οπότε έχουμε αυτό το πρωτόκολλο δράσης και έχουμε τα στελέχη του κόμματος που συνέχεια αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τη συμμετοχή τους στο πολιτικό γίνεστε, μέσα στο κόμμα. Ε, βέβαια, είπαμε ότι αυτά κατοχυρώνονται από τον ποινικό κώδικα, κάθε είδου βία ε, και έχουμε το πειθαρχικό όργανο του κόμματος που λαμβάνει μέτρα Οπότε είπαμε ότι έχουμε τα σχετικά σχέδια για την πολιτική βία, αλλά εγώ προσωπικά έφτιαξα ένα ad hoc πρωτόκολλο να είναι ένα εργαλείο και έτσι να μπορεί το κράτος να προστατεύσει τη γυναίκα σε δημόσιες θέσεις και γενικότερα όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα. Οπότε το επεξεργαζόμαστε αυτό, έχουμε μπλέξει και τον ΟΗΕ. Φέτος, φέτος όλα αυτά είναι ευκαιρία το 19 οπότε προχωρήσαμε και νομοθετικά πρόκειται για άλλο ένα είδος βίας γι' αυτό και χρειάζεται ειδική νομοθεσία όλες που είμαστε εδώ παρούσες ε, ασχολούμεθα με την πολιτική και οπότε θέλουμε να υπάρξει πρόοδος αυτά ευχαριστώ η Λορένα Μάτσεν. Ήδη σας το είπα στην αρχή και σε αυτό θα συνεχίσω. Το θέμα είναι το πώς η νομοθεσία θα γίνει πράξη. Άρα πρέπει να προβληθούν όλα αυτά προς τα έξω. Η πρόοδος και μέσα από την πρόοδο της τεχνολογίας. Τα δίκτυα, τα κοινωνικά, να τα προβάλλουμε όλα αυτά μέσα από εκεί. Και επίσης να αναλυφθεί δράση, όχι μόνο νομοθετική, θα πρέπει να δούμε πώς όλη αυτή η καινούργια οπτική για την ισότητα να είναι κάτι που διαπνέει πάσα πολιτική. Ως κοινωνίες, ως κράτη, να τα υλοποιήσουμε. Είναι κάτι σαν το κοινωνικό συμβόλαιο του κράτους με τους πολίτες, όχι μόνο εγώ με την νομοθεσία. Μπορεί να γίνει πρόοδος στην νομοθεσία, αλλά τι γίνεται στην πράξη. Θα πρέπει να συμβαδίζει η πραγματικότητα με την νομοθεσία. Αλλιώς δεν έχουν νόημα οι πρόοδοι, τα βήματα πρόοδου τέλο πάντων. Να τι πρέπει να κάνουμε οι γυναίκες. Και βοηθούν αυτές οι συνταλλαγές απόψεων. Εγώ προέρχομαι από την Παταγωνία της Αργεντινής και εκεί υπάρχουν ε, πάρα πολλά μέρη που είναι μακριά και δεν μπορούν να προβάλλουν ε, τον αγώνα αυτόν με τα κοινωνικά δίκτυα γιατί δεν έχουν ίντερνετ. Άρα θα πρέπει εμείς να πηγαίνουμε εκεί για να αναδείξουμε και εκείνες τις περιοχές. Έχουμε επίση την παρενόχληση για τι ε, ηθαγενείς γυναίκες που είναι απομονωμένε στον αγώνα αυτών, άρα θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, θα πρέπει να είμαστε δυναμικοί στις πολιτικές μας. Και άρα αυτό η διάσταση του φίλου να λαμβάνετε υπόψη από κάθε κυβερνητική απόφαση. Αύριο έχουμε ένα σημαντικό νομοσχέδιο για τις γυναίκες στην χώρα μας και γι' αυτό θα κατέβει ο κόσμος, θα πάει μπροστά στο κοινοβούλιο, θα διαδηλώσει και θα ε, ζητήσει να προχωρήσει η υπόθεση του νομοσχεδίου για την άμβλωση. Οπότε και εσείς μπορείτε να μας συμπαρασταθείτε, όπως είπα, με τα κοινωνικά δίκτυα. Από παντού, όλες οι γυναίκες. Στις 8.30 θα γίνει η διαδήλωση του συλλαλητήριων. Τώρα για την γυναικοκτονία. Κάθε 30 ώρες πεθαίνει μία. Νομοθετικά έχουμε κάνει βήματα πρόοδο. Αλλά για να προχωρήσουμε στο θέμα του mainstreaming χρειάζονται πόροι Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας από αυτή την άποψη. Και θα πρέπει οποιοδήποτε επιλήψιμη ανθρωποκτονία γυναίκας να θεωρείται γυναικοκτονία. Να είναι αυτό επιβαρυντική περίπτωση στη δίκη. να μην υπάρχουν ελαφρυντικά όταν έχουμε τέτοια ανθρωποκτονία. Συνεργασία για το μέλλον τώρα. Περισσότερη οργάνωση, περισσότερες τέτοιες μαζόξες, ανταλλαγή απόψεων, δικτύωση. Ε, οι δεσμοί απαραίτητοι ούτως ώστε παγκοσμίω να προβάλλουν τα δικαιώματά μας. Ε, Gabriela, Gabriela, παρακαλώ. Bueno, quería mm, Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να μιλήσουμε για την πολιτική βία. Καθότι η πολιτική ε, βία έχει προσθεθεί στην ε, βία κατά των γυναικών αναγνωρίστηκε ε, σε νομοθέτημα που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Και το, η, συνέλευση, η Βουλή ε, ασχολήθηκε με το θέμα. Υποβάλλονται δε ε, ολοκληρωμένα προγράμματα για την πολιτική κατά της βίας ε, και ειδικά κατά της βίας εναντίον στις γυναίκες που συμμετέχουν στην πολιτική, ε, τις γυναίκες που συμμετέχουν στα συνδικάτα, ε, στα, στις λέσχες, στις γειτονιές, στις κοινωνικές οργανώσεις κλπ. Και εμείς ζητούμε αυτό να θεωρείται ένα είδος πολιτικής βίας γιατί θέλουμε πραγματικά να συζητηθεί αυτός ο συνολικός νόμος έτσι ώστε να δημιουργηθούν εξειδικευμένα εργαλεία αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών στην ευρύτερη πολιτική. Επίσης αυτό που αναφερθήκατε στο ότι είμαστε ε, οι κόρες των λευκών μαντιλιών και οι μητέρες των πράσινων μαντιλιών. Ναι, εμείς θέλουμε ε, να ε, ε, ε, δημιουργήσουμε ε, αυτή την διασύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν, στο βίο παρελθόν, ανάμεσα στις γυναίκες που διαδήλωναν με τα λευκά μαντήλια στην πλατεία του Μαΐου, τις γυναίκες οι οποίες αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της δημιουργίας, για της δημοκρατίας, συγγνώμη, που αγωνίστηκαν για να έχουν πλέον ε, ε, να έχουν ε, την ευθύνη και την εξουσία πάνω στο σώμα τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο αγώνας που δίνουμε έτσι ώστε να γίνουμε κυρίαρχες των, του σώματός μας πρόκειται στην ουσία για αγώνα για την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Κοιτάξτε, εμείς ε, όλο το καλοκαίρι είχαμε πολύ, πολλές ε, συναντήσεις, ε, παρότι δεν δούλευε η Βουλή και είχαμε βεβαίως και τον πρόεδρο ο οποίος είπε ότι θα παρουσιάσει ε, το ε, σχέδιο για την ε, εθελοντική νόμιμη άμβλωση και μετά θα ξεκινήσει η, η συζήτηση σε επίπεδο κοινοβουλίου. Θα γίνουν λοιπόν οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις και ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του χρόνου θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά έτσι ώστε να υπάρξει η επικύρωση και φαντάζομαι ότι το Κοινοβούλιο ε, είναι αυτό το οποίο θα ε, ε, δώσει το τελικό πράσινο φως. Ξέρω ότι τα θέματα αυτά συζητιούνται για, και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως ας πούμε το θέμα της ενδιάμεσης μητέρας. Στην ε, ε, στην Αργεντινή συνήθως χρησιμοποιούμε τον όρο ε, αλληλέγγυα εγκυμοσύνη ή ενδιάμεση εγκυμοσύνη. Και οπωσδήποτε και εδώ όλα αυτά τα θέματα σχετίζονται με την επιβεβαίωση δικαιωμάτων και με την εμβάθυνση της ε, δημοκρατίας. Έχουμε μια ομάδα γυναικών ε, που προέρχονται από διάφορες πολιτικές ε, ομάδες και πλευρές που ακριβώς συζητούμε τα θέματα αυτά σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να μας βοηθήσετε σε αυτά τα σημαντικά θέματα τα οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε. κυρίως όσον αφορά αυτό το σχέδιο για την ε, εθελοντική νόμιμη άμβλωση. Κοιτάξτε, εσείς μπορείτε να δείξετε ενδιαφέρον, μπορείτε να μας υποστηρίξετε με οποιαδήποτε νομοθετική υποστήριξη από την πλευρά σας, ε, μέσω επιστολής, δηλαδή όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε εμείς που ασχολούμαστε, που συμμετέχουμε στην εκτελεστική ε, εξουσία αναγνώριση του αγώνα των γυναικών στην ε, Αργεντινή, ε, παρουσία όταν εμείς συζητούμε για αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά, σημαντικά όχι μονάχα στην Αργεντινή, αλλά και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, ε, μπορείτε να μας ε, παρακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε όταν η συζήτηση αυτή γίνει σε επίπεδο κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, ε, η κυρία Λόπες. Ευχαριστώ πολύ σε όλες ε, και σε όλους. Είσαστε λίγοι όπως ήθιστε, συνηθίζετε σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να καθίσουμε και να σκεφτούμε τα θέματα τα οποία αφορούν το, το, το, διαχωρισμό του φύλου και που αφορούν κυρίως τις γυναίκες, γιατί η πατριαρχία καλά κρατεί. Είναι προφανές ε, ότι υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο. Επίσης, πριν ε, μερικούς μήνες ξεκίνησε μια ιστορική συζήτηση και δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε η Σοφία, το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο εργασίας, το οποίο ε, ενεργοποιείται οποτεδήποτε, ε, οποτεδήποτε κάποιος ε, σύντροφος, άντρας ή γυναίκα αναφέρει παρενόχληση ή βία εργασιακή ε, μέσω ε, των ε, κοινωνικών δικτύων και λοιπά ξεκινάει μια διαδικασία γιατί όλοι ξέρουμε τις καταστάσεις. Επίσης υπάρχει μια ομάδα βουλευτριών που ασχολείται με εξειδικευμένα θέματα για την Νότια Αμερική για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που σε γενικές γραμμές ονομάζουμε λόγο ε, βίας μέσω των δικτύων κοινωνικής ε, δικτύωση. Αυτοί οι haters των κοινωνικών δικτύων ε, επιτίθενται πολύ ε, και με ιδιαίτερο τρόπο στις γυναίκες όπου αναφέρονται ας πούμε στα κοινωνικά δίκτυα για τις σεξουαλικές επιλογές, για τον τρόπο ζωής, πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την δημοκρατία. και οποτεδήποτε πιστεύω εγώ γίνεται μια προσπάθεια διεύρυνσης των δικαιωμάτων, οπωσδήποτε θα υπάρξει αντίδραση. Είναι η αντίδραση της Πατριαρχίας, είναι η αντίδραση ε, ε, του καπιταλισμού. Και επομένως ε, πραγματικά περιμένουμε τέτοιου είδους αντιδράσεις αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει πολιτική απόφαση όλων των πολιτικών ε, οργάνων έτσι ώστε να ε, δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην οικονομική, φυσική, σεξουαλική βία ε, την οποία υφίσταμεθα ως γυναίκες. Ε, είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου που αφορά ε, την ισοτιμία των ε, ευκαιριών, ίσες ευκαιρίες και θέλουμε πραγματικά και το Κοινοβούλιο ε, στην χώρα μου να αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο ένα εργαστήριο το οποίο όμως δεν θα παράγει μονάχα ε, λόγια ή ιδέες αλλά συγκεκριμένα μέτρα και ε, με τρόπο ώστε να υπάρχει δυνατότητα θεσμικής παρέμβασης όσον αφορά την ουσιαστική ισοτιμία, την ουσιαστική ισότητα. Ε, και οι νόμοι αυτοί πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Ε, θα πρέπει επίσης, όπως είπατε, ε, να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινότητας των αυτοχθόνων γυναικών. Στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκε ένα, μια ομάδα ε, που θα κάνουν 25 συνεδριάσεις σε δύο μήνες ε, ακριβώς ε, για γυναίκες ε, οι οποίες αντιμετωπίζουν και πιο εξειδικευμένα προβλήματα. Υπάρχουν πληθυσμοί για τις οποίες, όπως είναι ας πούμε οι αυτόχθονες γυναίκες, οι αγρότησες, οι γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο, που πρέπει να αντιμετωπιστούν με εξειδικευμένο τρόπο. Στην Αργεντινή δεν ε, συμβαίνει όπως σε άλλες χώρες Λατινικής Αμερικής όπου οι αυτόχθονες γυναίκες ε, έχουν ε, οργανωθεί. Στην Αργεντινή υπάρχουν ας πούμε οι πληθυσμοί Μαπούτσα, Σούι και λοιπά που πρέπει οπωσδήποτε να οργανωθούν διαφορετικά. Πρέπει πραγματικά να γίνει πολύ συγκεκριμένη εξειδικευμένη δουλειά με τις αυτόχθονες γυναίκες. Όσον αφορά τώρα το τι μπορεί να κάνει η Κοινοβουλευτική Ένωση, η παρακολούθηση μέσω των ε, δικτύων, κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στην ε, Αργεντινή, τι συμβαίνει στη Χιλή. Γιατί η παραβίαση των, των ε, δικαιωμάτων στη Λατινική Αμερική είναι κάτι συνηθισμένο ε, δεν πρόσεξαν το σημείο αυτό όλες οι κυβερνήσεις των χωρών. Γι' αυτό λοιπόν και στην Χιλή αποφάσισαν οι γυναίκες να κατεβούν στους δρόμους. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό που θα μπορούσε να γίνει ε, είναι το να παρακολουθείτε και μέσω συγκεκριμένης παρακολούθησης να ε, ε, ε, καθίσταται σαφής η παραβίαση που υφίστανται οι γυναίκες. Η Eurolat μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία. Οποιαδήποτε ευκαιρία δηλαδή δυνατότητας να γίνουν γνωστές περιπτώσεις, να αποκτήσουν ορατότητα περιπτώσεις γυναικών LGBT κλπ. που αντιμετωπίζουν ε, ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης ε, τα συστήματα μαθητείας που έχουν ξεχαστεί όσον αφορά αυτά τα, αυτές τις περιοχές. Επίσης, ε, οι γυναίκες πρέπει να δημιουργούμε δίκτυα γιατί ξέρουμε πώς να επιβιώνουμε εμάς ε, μας έχουν ε, μεγαλώσει με το να επαγρυπνούμε διαρκώς, να είμαστε σε μια κατάσταση επαγρύπνησης, γιατί πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά ε, και διαρκώς μαθαίνουμε να αποδεικνύουμε ας πούμε τι μπορούμε, τι είμαστε ικανές να κάνουμε. Εγώ Κοιτάξτε, δεν ε, θέλω να αναφερθώ και δεν στρέφομαι κατά ε, συντρόφων ή ανδρών. Απλώς θα πρέπει να αποδομηθεί ο, ε, αυτή η μορφή ε, πατριαρχίας και αυτή η μικροματσισμός όπως θα μπορούσα να τους ονομάσω. Και όταν σπάσουμε λοιπόν τα καλούπια και όταν σπάσουμε αυτές τις ε, εσφαλμένες μήτρες τότε θα έχουμε μια κοινωνία πιο πραγματική και πιο ε, δημοκρατική για όλες τις γυναίκες. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πολύ συγκινημένες που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τις αδερφές μας από την Ευρώπη και μακάρι να προχωρήσουν τα κοινωνικά μοντέλα και να μην έχουμε κι εμείς προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για ε, τα τελευταία πολύ θερμά σας λόγια. Ξέρω ότι είχατε κι άλλες ε, συνομιλίες εδώ πέρα. Εκμεταλλεύεστε την επίσκεψή σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ε, προσβλέπουμε στις μελλοντικές συναντήσεις σε άλλες περιστάσεις, στην Eurolat για παράδειγμα, αλλά και διμερός να σας ευχαριστήσω όλους. Καλό βράδυ σε όλους και θα τα πούμε σύντομα. This I finish, of course, uh, <laughs> Έτσι κλείνει και η σημερινή μας συνεδρίαση.